Uh, I would like to start the meeting. You might remember that we have uh, altered the agenda and... Το πρώτο θέμα για την απογευματινή ημερήσια διάταξη είναι η γνωμοδότηση Γκρομαντζόσκη για τις εκθέσεις 2012-2013 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Έγινε μια παρουσίαση της έκθεσης, υπήρξε μια συζήτηση μεταξύ των σκιωδών προθεσμία για τροπολογίες και σήμερα έχουμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Ο κύριος Γεζοντόφσκι θα πάρει το λόγο. Γεια σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που θεωρήσατε θετικά αυτό το σχέδιο. Σας ευχαριστώ για τις τροπολογίες και τα σχόλια τα οποία έχετε υποβάλει. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά να κάνω σήμερα, ειδικότερα. Θα ήθελα να σχολιάσω τις τροπολογίες, ομολογώ ότι υπάρχουν πολλές, 34 στον αριθμό. και θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους όσους έδειξαν ενδιαφέρον για το θέμα της επικουρικότητας και που υπέβαλαν αυτές τις τροπολογίες. Προσπάθησα να ξεχωρίσω αυτές τις τροπολογίες σε κάποιες κατηγορίες για να μπορέσουμε να είμαστε σαφέστεροι. Ήθελα λοιπόν να το μεθοδεύσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ξεχώρισα λοιπόν αυτές τις τροπολογίες σε ομάδες. Πρώτον, έχουμε τις τροπολογίες που προτείνουν νέες διατάξεις. Νέες διατάξεις έλεγα, αλλά βάσει υφιστάμενων κανονισμών ε, στις συνθήκες, διατάξεων στις συνθήκες. Ακόμη και βάσει των υφισταμένων γνωμοδοτήσεων. Παραδείγματο χάρη η τροπολογία Μπρέσο που θέλει τη συμμετοχή των τοπικών κοινοβούλιων ε, αναφέρεται σε αυτή την κατηγορία. Θα ήθελα λοιπόν ξεκινώντας να πω ότι πιστεύω ότι τέτοιου τύπου τροπολογίες μπορούν να προσθεθούν και με ενδιαφέρει να συμπεριλάβω αυτές τις τροπολογίες στην κοινοποδότηση. Μετά έχουμε τις εξειδικευόμενες τροπολογίες, μάλλον τροπολογίες εξειδίκευσης. Η υπαριθμόν 12 είναι μία, κύριου Πράγκελ, του κύριου η υπαριθμών 13. Είναι δηλαδή τροπολογίες οι, οποίοι, ε, οι οποίες εξειδικεύουν τον, έλεγχο, τον μηχανισμό ελέγχου σε σχέση με την επικουρικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καλό να περιλάβουμε αυτές τις τροπολογίες στη γνωμοδότηση. Αυτές λοιπόν θα μπορούσαμε να τις περιλάβουμε και αυτές στην τελική γνωμοδότηση. Τώρα περνάω στην τρίτη ομάδα. Μιλάω για τις τροπολογίες τώρα που εσωτερικά είναι ασυνεπείς. Αυτές είναι πρόβλημα. Είναι ασυνεπείς με τη γνωμοδότησή μου, αλλά και εσωτερικά αν θέλετε με τον εαυτό τους είναι ασυνεπείς αυτές τις τροπολογίες αν μπορώ να το πω έτσι. Αυτού του είδους οι τροπολογίες από τη μία πλευρά είναι απεσιόδοξες όσον αφορά τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων σε σχέση πάντα με την επικουρικότητα. Μιλάω για την τροπολογία 3 του κυρίου Κουρμπέτ. Αναφέρεται ειδικότερα ότι το γεγονός ότι οι διαδικασίες κίτρινης κάρτας και πορτοκαλί χρησιμοποιούνται σπάνια. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μια ολόκληρη σειρά από τροπολογίες που προσπαθούν να ενισχύσουν τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων ώστε να παίξουν σημαντικότερο ρόλο. Και εκεί έχουμε μια σύγκρουση όσον αφορά την προθεσμία δηλαδή το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα κοινοβούλια μπορούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους. Αυτό το οποίο πρότισα, πρότεινα και υποστηρίχθηκε και από κάποιους συναδέλφους και ενισχύθηκε μάλιστα ήταν να επιμηκύνουμε αυτήν την προθεσμία για την υποβολή γνωμοδετήσεων για νομοθετικές πράξεις. Δηλαδή θα ήθελα να το επεκτείνουμε πέραν των 8 εβδομάδων. Υπάρχουν τροπολογίε που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα επιμηκύνουν περαιτέρω. Αλλά υπάρχουν και κάποιες τροπολογίε που με σαφήνεια λένε ότι οι οκτώ εβδομάδες επαρκούν. Και τώρα όσον αφορά την σύγκρουση, αν θέλετε, των απόψεων, στην, στο σχέδιο γνωμοδότηση υπάρχει μια πρωτοβουλία για να ενισχυθεί η πρωτοβουλία των πολιτών χάρη στην οποία οι πολίτες μπορούν να παίξουν ένα μεγαλύτερο ρόλο στην Ευρώπη. Αυτό έχει περιληφθεί στο σχέδιο της γνωμοδότησης. Ανακεφαλαιώνω. Όταν πρόκειται για τις νέες τροπολογίες, οι οποίες καλύπτονται από το αρχικό σχέδιο της γνωμοδότησης, οκ, αλλά όταν μιλάμε για τροπολογίες εξειδίκευσης όπως τις αποκαλώ, νομίζω ότι υπάρχει ένας ρεαλιστικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή, θα σας υποβάλω συμβιβαστικές προτάσεις. Όταν πρόκειται για τις λιγότερο αμφισβητούμενες τροπολογίες, νομίζω ότι αυτές θα τις λύσουμε ψηφίζοντας. Η σύστασή μου είναι σαφής. Θέλω να ενισχύσω το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και θέλω να επιμικίνω την προθεσμία πέραν των 8 εβδομάδων και να υποστηρίξω την πρωτοβουλία των πολιτών. Τώρα, ένα άλλο θέμα που θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα συζήτησης είναι οι νέες λύσεις οι νέες λύσεις, οι οποίες είναι στο περιθώριο της συνθήκης, δηλαδή τροπολογία 18. Είναι η νομοθετική πρωτοβουλία για τα, εθνικό, ε, για εθνικά κοινοβούλια αποκαλείται πράσινη κάρτα. Ο κύριος Λάινεν έθεσε αυτό το θέμα πιο απαλά, παροτρύνοντας τα εθνικά και κοινοβούλια να συμμετάσχουν περισσότερο στη διαδικασία. Ευχαριστώ λοιπόν θα ακούσω πιο προσεκτικά τα έχετε να μας πείτε κύριε Λάινεν πάνω σε αυτό το θέμα διότι έχουν, έχουν σχέση με την έκθεση Μπροκ και Φερχόφστάτερ. Ε, και έχουμε και την τροπολογία 35 οι συνάδελφοι 25 μάλλον, με συγχωρείτε. Ε, οι συνάδελφοι προτείνουν την επισύναψη ενός ε, πρωτοκόλου στη συνθήκη κόκκινη και κίτρινη κάρτα για το Ευρωκοινοβούλιο και με αυτό το μηχανισμό το Ευρωκοινοβούλιο θα μπορεί να δεσμεύει τις πρωτοβουλίες που δεν ευθυγραμμίζονται με τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό όμως θα σήμαινε πολύ σημαντική μεταβολή της δομής μας και η τροπολογία 25 αν θέλετε συμβάλλει στην έκθεση Φερχόφστατερ. Σας υπενθυμίζω ότι επεξεργαζόμαστε την αρχή της επικουρικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, το 2000, για τα έτη 2012 13 και τα υπόλοιπα θα συμπεριληφθούν σε άλλες εκθέσεις. Από την άλλη πλευρά είμαι έτοιμος να περιλάβω συμβιβαστικές τροπολογίες στο σχέδιο της γνωμοδότησής μου και αναφέρομαι ειδικότητα στις τροπολογίες που δεν είναι συγκρουόμενες με τα υπόλοιπα. Αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων θα ψηφίσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ ο ε, από του ε, Λαϊκού Κομμάτου, ο κ. Πρέντα. Euh, Κυρία Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, σας ευχαριστώ για όλη την εργασία την οποία πραγματοποιήσατε. Δυστυχώς δεν είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απευθείας απόψεις πριν από σήμερα και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα με λίγα λόγια να εξηγήσω τα όσα υποκρύπτονται, αν θέλετε, κάτω από τις τροπολογίες τις οποίες πρότεινα. Ξεκινάω λέγοντας ότι κατά την άποψή μου ήταν σημαντικό να αναφερθούμε στον σεβασμό της αρχής της επικουρκότητας και της αναλογικότητας και να θυμίσουμε ότι δεν είναι μόνο τα εθνικά κοινοβούλια που είναι υπεύθυνα αλλά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να μην το ξεχνάμε αυτό. Συνεπώς, δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στο σημαντικό έργο βεβαίως των Εθνικών Κοινοβουλίων όσον αφορά την επαλήθευση ε, του σεβασμού των αρχών αυτών εκ μέρους ε, του Ευρωκοινοβουλίου, της Κομισιόν, ε, της Επιτροπής Περιφερειών. Αυτή είναι η γενική παρατήρηση που εμφανίζεται στις τροπολογίες μου 1, 5 και 13. Δηλαδή πρέπει να επαγρυπνούμε σε σχέση με τις αρχές. Και αυτό αναφέρεται και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όσον αφορά τώρα τη συμβολή των Εθνικών Κοινοβουλίων, μόλις αναφέρθηκα σε αυτήν, κατά την άποψή μου είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι το 2012 και το 2013 η διαδικασία της κίτρινης κάρτας ενεργοποιήθηκε. Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί σημαίνει ότι οι κανόνες που ισχύουν επιτρέπει τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στη λήψη αποφάσεων και ότι θέλουν και να συμμετάσχουν. Δεν υπάρχει δηλαδή μόνο ο κανόνος, κανόνας, αλλά υπάρχει και προσφυγή σε αυτόν τον κανόνα. Άρα ε, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι συνέβη αυτό, χρησιμοποιήθηκε ο μηχανισμός. Δεν μιλάμε για κάτι αόριστο δηλαδή, διαδικαστικό. Τώρα, όσον αφορά την επιμήκυνση της περίοδου των 8 εβδομάδων που είναι στη διάθεση των Εθνικών Κοινοβουλίων αυτή τη στιγμή, προσωπικά δεν θα σκοτωνόμουν την επιμικίνα. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τα εθνικά κοινοβούλια να εξοικειωθούν με τη διαδικασία, να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, προτού αξιολογήσουμε την ίδια τη λειτουργία και προβούμε σε μεταβολές. Μεταβολές που συνεπάγονται άλλωστε την τροποποίηση των συνθήκων. Γι' αυτό στην τροπολογία 15 ζητώ να σκεφτούμε το θέμα, αντί να προβούμε σε μία άμεση μεταβολή. Ίσως είναι σκόπιμο να περιμένουμε λίγο ακόμη, να συσσωρευτεί κάποια εμπειρία, να δούμε τις διάφορες πτυχές και να μην προτρέξουμε προς μία μεταβολή. Ε, μπορεί σε ένα-δύο χρόνια να αισθανθούμε ότι υπάρχουν άλλες αλλαγές που είναι αναγκαίες. Είναι πολύ πρόσφατη η διαδικασία για να προβούμε σε μεταρρύθμισή της και μια και αναφέρθηκα και στη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι απαραίτητη ώστε να προχωρήσουμε στον έλεγχο της επικουρκότητας στην πλήρη ανάπτυξή του. Χρειαζόμαστε λοιπόν συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να αναφέρεται και στην πρακτική της εξέταξης της επικουρικότητας από τα Εθνικά Κοινοβούλια διότι υπάρχουν σημαντικές αποκλήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση αυτών των δύο αρχών. Δεν έχουμε ενότητα στην αντίληψη όσον αφορά την εξέταση των πρακτικών. Τι είναι σωστό και τι είναι δηλαδή. Πάντα σε σχέση με την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Συνεπώς, οι αρχές αξιολόγησης δεν πιστεύω ότι πρέπει να επιβληθούν εκ των άνω από τους θεσμούς, διότι θα διαφεύγαμε από το πνεύμα το νομοθετικό, το πραγματικό της ουσίας. Αφήσουμε, ας αφήσουμε λοιπόν τα κοινοβούλια να λειτουργήσουν. Ας τα ενθαρρύνουμε να προχωρήσουν για να δούμε πώς μία τέτοια αλληλοεπίδραση μπορεί να μεθοδευτεί και να αξιολογηθεί. Δεν πιστεύω ότι κατά τρόπο προπέτη πρέπει αυτή τη στιγμή να προσπαθήσουμε να δώσουμε ήδη μαθήματα αν θέλετε. Πρέπει να συνεργαστούμε μέσα στο πλαίσιο της επικορικότητας. Προτείνω όπως και άλλοι συνάδελφοι την κατάργηση του άρθρου για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών γιατί δεν πιστεύω ότι έχει θέση εδώ στην έκθεση επικουρικότητας. Ο κύριος Σουζαντόφσκι ήδη αναφέρθηκε σε αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ο Σαλ Κέρενς για τους φιλελεύθερους όχι εσείς. Η κυρία, μάλιστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε λίγο διεξοδικότερα αυτό το ζήτημα γιατί θα πρέπει βέβαια να επιτύχουμε μια πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων και της Εθνικής Αρμοδιότητας αφενός ε, και του των δικών μα αρμοδιοτήτων ω Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου και ε, κατά συνέπεια θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα αυτό το ζήτημα ε, και με προσεπτικό τρόπο να ε, προτείνουμε ότι θέλουμε να γίνει περαιτέρω δουλειά σε σχέση με αυτό το ζήτημα γιατί βέβαια το, το, το ότι θα κάνουμε θα έχει και ένα αντίκτυπο ντόμινο αν θέλετε και σε άλλες δηλαδή επιτροπές και σε άλλες αρμοδιότητες κοινέ που έχουμε στο επίπεδο δηλαδή της Ευρώπης. Ε, κατά συνέπεια θεωρούμε πως η τροπολογία 25 είναι ιδιαίτερα σημαντική, έχει νόημα δηλαδή σε ό,τι αφορά τα εθνικά κοινοβούλια και νομίζω πως ε, θα έχουμε και τη δυνατότητα να εξετάσουμε και από πολιτικής και από τεχνικής ε, άποψης ε, το ζήτημα του κατά πόσο θα πρέπει να επεκταθεί όχι η προθεσμία των 8 εβδομάδων. Ε, εμείς ε, τουλάχιστον δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει ε, να επεκταθεί η φυστάμενη προθεσμία των 8 εβδομάδων μέχρι τουλάχιστον να δούμε αν αξιοποιείται ή όχι από το Εθνικά Κοινοβούλιο το νέο εργαλείο καθώς είναι πραγματικά πολύ καινούριο και δεν έχουμε ακόμα δει να χρησιμοποιείται εκτεταμένα από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πάντως πρόκειται επαναλαμβάνω για μια λεπτή ισορροπία γιατί πρέπει να επιτύχουμε πολιτική βούληση από τη δική μας πλευρά και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα εθνικά κοινοβούλια, στο εθνικό δηλαδή επίπεδο. Οτιδήποτε δηλαδή εμείς ε, θα κάνουμε από την πλευρά μας θα πρέπει ε, να ε, αποφύγει οποιαδήποτε πολιτική κρίση στην Ευρώπη για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε, ο κύριος Σόπφλιν. Ευχαριστώ. Και πρόεδρε και ευχαριστώ κύριο Αντοσίου για αυτήν την έκθεση. Είναι κάποιες τώρα από τις σκέψεις που έκανα, ακούγοντας τα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα, είναι ότι η αίσθηση που έχω ότι η προθεσμία των 8 εβδομάδων για την ε, έκφραση αιτιολογημένη γνώμη από την πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων πραγματικά αποτελεί μια στενή προθεσμία. Δηλαδή θα πρέπει να του δοθεί περισσότερο χρόνο στα Εθνικά Κοινοβούλια να εκφράζονται. Και το γεγονό ότι δεν έχουμε λάβει πολλέ από αυτέ από την πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων, πράγματι μα παραπέμπει ότι πρέπει, θα πρέπει να γίνει κάποια παραπάνω σκέψη. Εκείνο πάντω που σκέφτομαι είναι ότι είναι ότι εμείς εξετάζουμε ένα ε, ολόκληρο ευρωπαϊκό αν θέλετε ε, πλαίσιο και από εκεί και ε, η ιεραρχία σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι εμείς βρισκόμαστε πάνω-πάνω από εκεί και μετά είναι τα Εθνικά Κοινοβούλια, Περιφερειακές Αρχές και Κοινοβούλια και μετά οι ίδιοι οι πολίτες. Οπότε θα ήθελα εγώ να προσπαθήσετε να επιτύχετε έναν δεσμό ανάμεσα σε εμά, απευθεία δεσμό και στους πολίτες δηλαδή να εκφράσουμε ότι οι πολίτες ε, είναι θεμητό να και θα πρέπει να περιλαμβάνονται ε, μέσα στο ε, επίπεδο της πολιτικής δράσης, τη επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε δηλαδή πως οι κανονικές διαβουλεύσεις όπως αυτές λαμβάνουν χώρα δεν αποτελούν εμπόδιο, αντιθέτως είναι χρήσιμες και, και σε ό,τι αφορά ε, κάποιες από τις τροπολογίες τώρα οι οποίες ε, προτάθηκαν ε, και ειδικότερα αναφορές που γίνονται στο Green Castle President Card θεωρώ ε, πως ε, πραγματικά θα δημιουργήσουν σύγχυση σε ό,τι αφορά ακριβώς την οριζόντια και κάθε τη δομή που έχουμε στο πολιτικό πεδίο. Κατά συνέπεια δεν είμαι σίγουρος εάν αυτές οι προτάσεις για συμπερίληψη της πρωτοβουλίας της Πράσινης Κάρτας είναι επιθυμητές. Τελικά το ερώτημα είναι ε, κατά πόσο θέλουμε να αποδεχτούμε οποιαδήποτε πρόταση η οποία μας καλεί να προβούμε σε ε, τροποποίηση της ε, συνθήκης. Έχουμε και την έκθεση του Σάλλου Βερχόφσταντ που θα συζητηθεί και πάλι το ίδιο ζήτημα, δηλαδή κατά πόσο χρειάζεται τροποποίηση της συνθήκης. Κάποιοι λένε ότι αποκλείεται, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε, άλλοι λένε ναι, πως είναι χρήσιμο, θα πρέπει να το κάνουμε. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, πάντως η Green Card, η πράσινη κάρτα κατά τη δική μου άποψη σίγουρα προϋποθέτει τροποποίηση της συνθήκης και κατά συνέπεια δεν νομίζω πως πρόκειται για μια χρήσιμη πρόταση. Ευχαριστώ λοιπόν τον συγκεκριτή για την εργασία του και αυτά από την πλευρά μου. Ο Ρίσαρτ Κόρμπιτ έχει τώρα το λόγο. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγκεκριτή για τη δουλειά που έχει κάνει. Να θέσω και εγώ κάποια σημεία. Καταρχήν, ε, σε ό,τι αφορά την προθεσμία των 8 εβδομάδων, και εγώ θεωρώ πω ε, δεν αποτελεί ένα ενδεδειγμένο χρονικό πλαίσιο ε, προκειμένου να προβούμε, για παράδειγμα, σε μετροποίηση τη συνθήκη. Χωρί να περιορίζομαι δηλαδή μόνο σε αυτό το σημείο. Στην τοπολογία μου παριθμών 17 υπάρχει μια σχετική αναφορά Αναφέρεται δηλαδή εκεί ότι η εν λόγω προθεσμία θα πρέπει να τη χάνει μια ευέλικτη ερμηνεία. Ε, για παράδειγμα, ε, υπάρχει για ένα προηγούμενο σε ό,τι αφορά τι προθεσμίε ε, στο πλαίσιο τη δεύτερη εναού, δηλαδή 6 και μετά 8 εβδομάδε. Έχουμε δηλαδή κάποιε συμφωνίε τι οποίε έχουμε επιτύχει με την Επιτροπή ότι δεν ξεκινάει δηλαδή με επίσημη υποβολή από την πλευρά της Επιτροπής σε μια διαδικασία σε περίπτωση που δεν έχουμε εκπληρώσει την σχετική προθεσμία όταν πρόκειται ε, για επικείμενες διακοπές ε, Πάσχα ή Χριστουγέννων. Οπότε ενδεχομένως μια χρήσιμη ιδέα θα ήταν μια εκ των προτέρων υποβολή ενός ε, κειμένου χωρίς δηλαδή να, να προηγείται αυτή η ανεπίσημη της επίσημης υποβολής μιας πρότασης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια να τηρούν ε, τη συγκεκριμένη προθεσμία χωρίς ταυτόχρονα να χρειαστεί η τροποποίηση της συνθήκης. Από εκεί και μετά, συμφωνώ και με άλλους ε, προαλήσαντες ότι δηλαδή η παράγραφος ότι αφορά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται όπως είπατε και εσείς ε, κύριε Σιγητά η τροπολογία 25 αναφέρεται περισσότερο στην έκθεση Verhofstadt και αναφορά στην έκθεση πρωτοβουλία πολιτών είναι το κατάλληλο σημείο που θα πρέπει να περιληφθεί. Κύριο Σέφλιν δηλαδή. ε, ένα τρίτο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω. Η επικοινωνικότητα δεν αποτελεί στην πράξη, τουλάχιστον όχι συχνά, ένα πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή η κίτρινη ε, κάρτα με την απαραίτητη πλειοψηφία έχει ενεργοποιηθεί, έχει δηλαδή αξιοποιηθεί δύο φορές μέσα στα τελευταία έξι χρόνια και νομίζω πως υπάρχουν μια σειρά από λόγοι που, στους οποίους οφείλεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή οι ε, νομοθετικές ε, ε, τροποποιήσεις αφορούν υφιστάμενη νομοθεσία συχνά, ε, είναι γνωστές οι διαδικασίες που ακολουθούμε. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από λόγου που δεν αξιοποιείται αυτή η διαδικασία. Τα εθνικά κοινοβούλια προφανώ ενδιαφέρονται για προτάσεις αλλά ε, ε, αυτό που μας ενδιαφέρει τελικά είναι η ουσία της αναλογικότητας. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ ε, προτείνω μιας, κάποιες τροπολογίες οι οποίες λένε ότι δεν θέλουμε να περιχαρακωθούν σε ένα ρόλο δηλαδή ελέγχου της επικορικότητας στα Εθνικά Κοινοβούλια και τίποτα πέρα από αυτό. Αυτό που λένε οι δικές μου τροπολογίες είναι ας ε, πούμε κάτι ευρύτερο, κάτι δηλαδή περαιτέρω επί της ουσίας. Ε, και γι' αυτό για παράδειγμα χαιρετίζουμε την ε, πρωτοβουλία Παρός δηλαδή σε ό,τι αφορά τις ε, προτάσεις τροποποιήσεων που μπορούν να κάνουν τα Εθνικά Κοινοβούλια απευθεία στην Επιτροπή. Όμως το κυρίως όχημα, αν θέλετε ο κύριος Διάβλος για να τροποποιήσει την λήψη πολιτικών αποφάσεων είναι ο Υπουργός που εκπροσωπεί την εκάστοτε χώρα στο Συμβούλιο. Γιατί βέβαια αυτός ο Υπουργός εκπροσωπεί το Εθνικό Κοινοβούλιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο Συμβουλίου. Αν λοιπόν υπάρχει μια πρόσκληση, για παράδειγμα, ε, να μιλήσει σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή ο Υπουργό, ο οποίο θα βρεθεί ε, την επόμενη εβδομάδα σε ένα συμβούλιο, ε, τότε δίνεται ακριβώ τη δυνατότητα στο Εθνικό Κοινοβούλιο να επηρεάσουν την λήψη των πολιτικών αποφάσεων επί τη ουσία. Δηλαδή υπάρχει και η εθνική εκπροσώπηση μέσω του Υπουργού και ε, προφανώς οποιαδήποτε κίνηση προς την ενδυνάμωση του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων έναντι του Υπουργού του είναι επιθυμητή και ε, από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά την προθεσμία των τροπολογιών θα ενημερώσω τη γραμματεία γιατί ενδεχομένω θα ήθελα να υποβάλω κάτι ακόμα. Δεν ξέρω αν ε, ε, θέλει κάποιο άλλο να πάρει το λόγο, λέει ο Πρόεδρο. Παρακαλώ. Thank you. I too would like... Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή με τη σειρά μου. Βασικά πρέπει να πω ότι συμφωνώ με αυτή την εισήγηση. και πιστεύω ότι η περίοδος των 8 εβδομάδων δεν είναι επαρκής. Διαβάζοντας λοιπόν όλες τις τροπολογίες τρόπον την Α, θα ήθελα να είχα σκεφτεί την, την ιδέα να υποβάλω προτάσεις για να λύσουμε τα προβλήματα του ελέγχου της επικουρικότητας χαμηλώνοντας το σημείο εκκίνησης. Βεβαίως όλα αυτά συνεπάγονται με τα πολύ των συνθήκων και αυτό θα γίνει ακόμη πιο σημαντικό όταν θα φτάσουμε στο να θέλουμε να υποκινήσουμε τα εθνικά κοινοβούλια να προχωρήσουν σε έλεγχο των, της επικουρικότητας. Γιατί αυτή τη στιγμή κάποια κοινοβούλια το πράττουν, πράττουν τον έλεγχο δηλαδή, και άλλα κοινοβούλια δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Εάν ε, ήταν ευκολότερο να λειτουργήσει η κίτρινη κάρτα, τότε θα υπήρχε και κίνητρο για τα κοινοβούλια να το εφαρμόσουν. Όμως, ίσως αν θέλετε αυτό το θέμα ξεπερνάει το θέμα που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή την έκθεση του 12 και του 13. Μ' άρεσε λοιπόν η πρόταση που έκανε ο κύριος Κόρπ όσον αφορά την ευέλικτη ερμηνεία της περίοδου των 8 εβδομάδων. Μεταβάλλοντας τη ουσία, την ουσία χωρίς να μεταβάλουμε τις συνθήκες είναι πάντοτε ενδιαφέρον. Έχουμε δύο τροπολογίες που δεν νομίζω ότι αμφισβητούνται από τους πράσινους. Ελπίζω να μπουν στο τελικό κείμενο και έχω και μία ερώτηση όσον αφορά την 25 σε σχέση με την κόκκινη και την κίτρινη κάρτα. Δηλαδή κατά πόσο το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει σχετικό έτοιμο στα εθνικά κοινοβούλια. Αναρωτιέμαι εάν οι συντάκτες της πρότασης σκέφτηκαν πόσο προσωπικό χρειάζεται. Ε, έχουν κάνει δηλαδή κάποια προκαταρτική αξιολόγηση του κόστους ώστε να ξέρουμε πόσα χρήματα απαιτούνται για να γίνει σωστά αυτή η δουλειά. Σας ευχαριστώ. Ραμάν Χαραλή. Θα ήθελα και εγώ να συμβάλλω στη συζήτηση. Ειδικότερα θα ήθελα να σας πω πώς βλέπω τα πράγματα. Τα τρία τελευταία χρόνια Ε, ε, ήμουν βουλευτής στην Ισπανία και συνεπώς ξέρω τα προβλήματα από αυτή την πλευρά. Έχουμε μικτές επιτροπές των δύο σωμάτων ε, των κοινοβουλευτικών της Ισπανίας και κάθε εβδομάδα ανασκοπούμε τα διάφορα θέματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει φυσιολογικά, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή δεν απαιτείται να μπει κανείς ε, στις λεπτομέρειες, στις προθεσμίες, να υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της επικουρικότητας. Η επικουρικότητα είναι μια αρχή ε, της συνθήκης της Λισαβόνας και όπως τα έλεγε ο Ρίτσορτ Κόβερτ, ε, δεν δημιουργεί κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα διότι η Κομισιόν είναι πολύ προσεκτική, ξέρει ακριβώς μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πού δεν πρέπει να πατήσει. Ο αντιπρόεδρος Τίμερμαν μας είπε ότι είχε την πρόθεση να ξεκινήσει μία συζήτηση ώστε οι πρωτοβουλίες της Κομισιόν να μην παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας. Θα ήθελα λοιπόν να πω στον εισηγητή ότι δεν συμμερίζομαι την προσέγγιση του, τη στενή, τη στενάχωρη αν μπορώ να την πω έτσι ότι απόλυτα πρέπει να εφαρμόσουμε την επικουρικότητα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με την επικουρικότητα, τολμώ να πω. στην ομάδα μου ε, μπορώ να ισχυριστώ ότι συμφωνούμε με τις τροπολογίες του Ρίτσαρντ. Ε, δεν χρειάζεται να φτιάξουμε ολόκληρο αμυντικό σύστημα για να υποστηρίξουμε την αρχή της επικουρικότητας. Είναι στην, στη συνθήκη της Λισαβόνας εφαρμόζεται, χρειάζονται άραγε ε, μεγαλύτερες προθεσμίες. Όχι. Έρχομαι από μια χώρα που έχει τις περιφέρειες με ενισχυμένες εξουσίες, ούτε τα λέντερ της Γερμανίας δεν έχουν τόσες αρμοδιότητες και εξουσίες. Και μπορώ να σας πω ότι μέσα στις 8 εβδομάδες η Αυτόνομη Επιτροπή στην Ισπανία μπορεί να γνωμοδοτήσει. Όταν λοιπόν υπάρχει μια αίσθηση παραβίασης της αναλογικότητας ή της επικορικότητας εξετάζεται η έκθεση της Αυτόνομης Επιτροπής από το Κοινοβούλιο και απευθύνει το σχετικό διάβημα στις Βρυξέλλες. Τη σχετική έκθεση μάλλον. Ε, δεν νομίζω ότι αξίζει να διαμαρτυρόμαστε και να γκρινιάζουμε ότι δήθεν δήθεν δεν υπάρχουν αρχές για την αξιολόγηση της επικουρικότητας. Πολλά πράγματα έχουμε, έχουμε πολλές παραμέτρους, δεν ζητάμε τη σελήνη. Λοιπόν, είμαι αντίθετος με αυτό το πνεύμα. Το αρνητικό εννοώ, το οποίο αναδύεται από αυτή την έκθεση. Θα βρούμε τρόπους συμφωνίας. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι η επικουρικότητα καταρχήν είναι σημαντικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 21ου αιώνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και δεν βλέπω γιατί πρέπει να επιμηκυνθούν οι προθεσμίες, διότι τελικά όλη η νομοθετική διεργασία της Ένωσης θα υπονομευτεί. Σας το λέω με σαφήνεια γιατί έτσι πιστεύω. Ε, Αρχικά είχα πει ότι δεν θα πάρω το λόγο, λέει ο επόμενο ομιλητή, αλλά μετά το συνάδελφο Κόρμπετ θα ήθελα να παρέμβω σε ένα σημαντικό σημείο. Σωστά υπογράμμισε ότι ο έλεγχο τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα είναι μία πτυχή. Το Υπάρχει και ένα βαθύτερο πρόβλημα. Το είχα ε, εξετάσει πριν από 15 χρόνια μετά από αίτημα του Γιούγκερ που μου ζήτησε να συντάξουμε μία έκθεση σε σχέση πώς, του πώς θα μπορούσαν να συμμετέχουν περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια στο νομοθετικό έργο της Ένωσης. Καταλήξαμε λοιπόν τότε στο συμπέρασμα ότι τα ε, κοινοβούλια συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Αυτά που ξεκινούνται πιο νωρίτερα επηρεάζουν ε, και τα αποτελέσματα. Το Folketing της Δανίας ήταν ο πρωταθλητής. Έχει μία κουλτούρα που αν θέλετε οφείλεται στο ότι συχνά έχουν κυβερνήσεις μειοψηφίες. Επειδή δε οι κυβερνήσεις είναι μειοψηφίες, πρέπει να υποστηρίζεται παρόλα αυτά από μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία και έτσι το Folketing συμμετείχε περισσότερο στην όλη διαργασία των υποθέσεων του κράτους. Ακόμη τα κείμενα επικυρώνονται εθνικά αν συμμετάσχουν εξ αρχή τα κοινοβούλια. Τότε λοιπόν αυτή η διαδικασία ε, από τότε αυτή η διαδικασία μοιάζει να εξαφανίστηκε. Έχουμε ακροάσεις στα Συμβούλια των Υπουργών και πριν από την υποβολή ενός νομοθετικού κειμένου η Κομισιόν αναζητεί τα σχόλια των κρατών μελών μέσα στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Συμβουλίου των Υπουργών. Παραδείγματο χάρη πήγαινα στο Συμβούλιο του Περιβάλλοντο στην εποχή εκείνη, αυτό γινόταν τακτικότατα. Ήταν ανοιχτή η συζήτηση. Αυτοί λοιπόν που θέλανε να έχουν μια αντίληψη πώ ε, γίνεται κατανοητό το κείμενο ε, στο προσχέδιό του, είχαν τη δυνατότητα να δούνε αν το κείμενο το προτινόμενο είχε πιθανότητες να περάσει τα σύνορα αν θέλετε, να προχωρήσει δηλαδή. Ε, ε, ε, σε όλα τα κοινοβούλια θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική μία επεξηγηματική σημείωση της κυβέρνησης που να εξηγεί ποιε είναι οι συνέπειες, ο αντίκτυπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη και έτσι θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε πώς κατανοούν τα νομοθετικά κείμενα οι κυβερνήσεις διότι έχουμε μία γλώσσα που χρησιμοποιείται στις Βρυξέλλες και μία διαφορετική κατανόηση στα κράτη-μέλη. Όλα αυτά τα σημεία συνεπώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν κάπου την συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων με την έννοια που σκιαγράφησε ο Ρίτσαρτ. Είναι θλιβερό να διαπιστώνουμε το υψηλό ή το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των μεν και των δε. Μιλάω πάντοτε για τα εθνικά κοινοβούλια. Υπάρχουν κάποιοι που έρχονται εδώ με πάθος και γνώση και υπάρχουν άλλοι που δεν τους ακούμε και ποτέ. Λοιπόν, αν θέλουμε να εμβαθύνουμε, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτά τα αρχικά και μπορώ να αναζητήσω αυτή την έκθεση που είχα συντάξει πριν από τόσα χρόνια που σας έλεγα και να τη δώσω στη γραμματεία. Σας ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο θα δώσει και πάρει το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Ευχαριστώ. Ε, όλους τους ε, ομιλητές ε, για όλη τη συζήτηση που κάναμε εδώ. Θα ήθελα να κάνω και κάποια σχόλια από την πλευρά μου. Καταρχήν ε, υπάρχουν κάποιες από αυτές τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί που θα τις ονόμαζα διευκρινιστικές και θα μπορούσαν πράγματι να προσθεθούν στην έκθεσή μου και δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Για παράδειγμα αναφέρομαι εδώ στις τροπολογίες 1, 5 και 13 από τον κύριο Πρέντα δηλαδή. Γιατί, Γιατί εν λόγω τροπολογίε ουσιαστικά αποσαφηνίζουν τα όσα ήδη περιλαμβάνονται στη δική μου, στο δικό μου σχέδιο έκθεση. Σχέδιο Ε, μετά, σε ό,τι αφορά την προθεσμία των 8 εβδομάδων, θα προετοιμάσω ε, μια συμβαστική διατύπωση, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω με ένα κείμενο που θα λέει ότι 8 εβδομάδες επαρκούν ως προθεσμία. 8 εβδομάδες για μία γνωμοδότηση στο πλαίσιο νομοθετικής διαδικασίας δεν υπάρχει. Δηλαδή μια νομοθετική διαδικασία εδώ στις Βρυξέλλες μπορεί να διαρκέσει τρία χρόνια στο πλαισιο νομοθετικης διαδικασιας δεν υπαρχει δηλαδη μια νομοθετικη διαδικασια εδω στις βρυξελλες μπορει να διαρκεσει 3 χρονια στο συνολο της. Και συμβαίνει συχνά να διαρκέσει τόσο πολύ. Οπότε 8 εβδομάδες ως προθεσμία για την διαμόρφωση μιας γνώμη στο πλαίσιο μιας ε, διαδικασίας η οποία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα δεν ε, είναι ενδεδειγμένο. Δηλαδή δεν υπάρχει μια τέτοια προθεσμία για ε, τα εθνικά κοινοβούλια, τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια και κατά συνέπεια τα αποθαρρύνει από μια συμμετοχή. Ε, και θα ήθελα εδώ να λάβετε υπόψη σας ότι μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή ζητάμε από τα εθνικά κοινοβούλια να τοποθετηθούν με γνωμοδοτήσεις για πολύ συγκεκριμένα θέματα. Οπότε ο προσανατολισμός που θα ήθελα να ακολουθήσουμε είναι ε, να υπάρχει μια περισσότερη ευελιξία. Όχι λοιπόν να αξιώσουμε μια παράταση της προθεσμίας ε, προκειμένου ε, και προκειμένου να γίνει αυτό να υπάρξει και μια τροποποίηση της συνθήκης μια ευέλικτη προσέγγιση θέλουμε και κατά συνέπεια ευέλικτη και διατύπωση της γνωμοδότησης. Τώρα, ε, ε, σε ό,τι αφορά την ε, τροπολογία για νομοθετική πρωτοβουλία από την πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων, μου δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Και αυτό γιατί, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο που συνοδεύει τη συνθήκη τη Λισαβόνα και υπήρξαν πολύ συγκεκριμένε προποθέσει για τη διατύπωση του εν λόγω πρωτοκόλλου. Γιατί τα εθνικά κοινοβούλια χρησιμοποιούν την αρχή της επικουρικότητας. Γιατί ε, καλούνται να τοποθετηθούν με γνωμοδοτήσεις επί κανονισμών. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει διοικητικού χαρακτήρα αποφάσεις οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην εθνική νομοθεσία. Ε, εκεί λοιπόν τοποθετούνται με γνωμοδότηση τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αντιθέτως στις οδηγίες καλούνται τα Εθνικά Κοινοβούλια να εφαρμόσουν στην πράξη και να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τα όσα περιλαμβάνονται εν ίδια στην οδηγία. Άρα λοιπόν κατά τη δική μου άποψη η αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται ακριβώς στο πλαίσιο αυτών των ε, οδηγιών και των ε, κανονισμών. Και από εκεί και μετά η πρωτοβουλία η νομοθετική, ε, νομίζω πως εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε τα όσα είπε ο κύριος Κορμπέντ. Δηλαδή μιλάμε για κοινοβουλευτική πλειοψηφία που αποτελεί την την, ε, τον νόμο και τον κανόνα σε όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή εφόσον συγκεντρώνεται πλειοψηφία υπέρ ενός αιτήματος σε ένα εθνικό κοινοβούλιο, εκείνο που θα πρέπει να κάνει το λόγο κοινοβούλιο είναι να ενθαρρύνει την κυβέρνηση προκειμένου να υποθέσει μια νομοθετική πρόταση που θα υποβληθεί στο, στο Συμβούλιο. Άρα λοιπόν πραγματικά θα είμαι πολύ προσεκτικό και επιφυλακτικό σε ό,τι αφορά αυτή την τροπολογία των πρασίνων. Πάντω, σε ό,τι αφορά την προθεσμία των 8 εβδομάδων, θα είμαι πιο ευέλικτο και πιο μαλακό εντό εισαγωγικών. Αυτά. Στι 5 Μαου, λέει ο ε, Πρόεδρο, θα ψηφίσουμε επ' αυτή τη ε, γνωμοδότηση. Ε, περνάμε λοιπόν στο σημείο 11 τη ημέρα σα διάταξη συζητήσει ο κύριο Σόπλιν σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Έχουμε λοιπόν μια δεύτερη συζήτηση και θα θέσουμε και ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ο λόγος λοιπόν στον Γιώργο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι μόλις έλαβα αυτό το το κείμενο δηλαδή της εμπειρίας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών κατά τρία ε, πρώτα χρόνια. Δεν είχα αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου για να το διαβάσω, αλλά πραγματικά δείχνει να είναι μια πολύ χρήσιμη ε, σύνοψη. Θα ήθελα να κάνω λοιπόν κάποιες, ε, κάποια γενικά σχόλια. Καταρχήν να πω ότι έχει υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών από την πλευρά λοιπόν της, της κοινωνίας των πολιτών, ε, ε, όχι από όλη την κοινωνία των πολιτών, αλλά πάρα πολλές ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν εμπλακεί εδώ στο lobbying, στην ανταλλαγή απόψεων. Ε, δύο ακροάσεις ε, θα έχουμε και εδώ στην δική μας Επιτροπή και σε μια ακόμα κοινοβουλευτική επιτροπή. Ε, υπήρξε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολλά email λάβαμε, οπότε συγκεντρώνει λοιπόν αυτό το ζήτημα πραγματικά το ενδιαφέρον του κοινού και βέβαια, ε, κατά συνέπεια, καθίσταται και από πολιτική άποψη πολύ σημαντικό. Και αυτό γιατί, εάν ε, δούμε ε, την, την πόσο, πόσο μακρο, αν θέλετε, η χρονοβόρα ήταν η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα καταλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι να εμπλέξουμε εδώ και την ε, κοινωνία των πολιτών. Και βέβαια ε, η προσθήκη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών δεν ε, επαρκεί από μόνη της. Χρειάζεται πολιτική βούληση και η πολιτική βούληση συνεπάγεται βέβαια και μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων φορέων. Και εδώ μιλάμε κράτη-μέλη, Συμβούλιο, Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια και η κοινή γνώμη δηλαδή με άλλα λόγια οι ίδιοι πολίτες. Έτσι λοιπόν ο πολίτης, ο Ευρωπαίος πολίτης παραμένει αδύναμος αν θέλετε στο πλαίσιο αυτού του οικοδομήματος. Μόνο μια μικρή μειοψηφία των 500.000 Ευρωπαίων ε, πολιτών θεωρεί τον εαυτό του ως ε, τέτοιο πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα θυμόσαστε και το Ιρλανδικό δημοψήφισμα που έδωσε, μας έδωσε και αυτό το νέο όρο του disconnect, δηλαδή όπου κανείς ε, ναι μπορεί εύκολα να νιώσει ως πολίτης της Ιρλανδίας αλλά όταν χρειάζεται να ψηφίσει ενός ευρωπαϊκού ζητήματος δεν νιώθει αυτή την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Και εδώ λοιπόν είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά την ε, διαδικασία της ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης και εδώ έχει να παίξει το δικό της ρόλο η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών. Μπορεί δηλαδή να επιφέρει σημαντικές αλλαγές εντατικοποιώντας ακριβώς την ταύτιση του πολίτη με ε, την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και εάν μια ε, πρωτοβουλία πολιτών Ε, υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος αυτή η ταύτιση να μετατραπεί σε αδιαφορία ή ε, στη χειρότερη περίπτωση σε εχθρότητα. Τώρα θα ήθελα να τονίσω εδώ πως η πρωτοβουλία αυτή είναι και νομικό και ε, πολιτικό ε, εργαλείο. Η νομική πτυχή προφανώς είναι εμφανής, αλλά η πολιτική ενδεχομένως να μην είναι πολύ εμφανής. Και κάναμε και μια συζήτηση μόλις τώρα και με τον κύριο Κόρμπετ δηλαδή. Ε, κινητοποιεί τους Ευρωπαίους ε, πολίτες. Ναι, εντάξει δεν κινητοποιεί πάρα πολλά εκατομμύρια, αλλά ναι. 6 εκατομμύρια μέχρι στιγμής έχουν εμπλακεί στο σύνολο των 50 ε, ενός πρωτοβουλειών πολιτών. 51 πρωτοβουλίων πολιτών που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα. Και ε, ε, αυτό το εργαλείο εφόσον λειτουργεί σωστά μπορεί να ε, μεταφέρει περισσότερη ισχύ, περισσότερη δύναμη στους ίδιους τους πολίτες καθώς έχει συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής αυτή η ισχύ εδώ στις και επειδή αυτό το νέο εργαλείο, αυτό το νέο σύστημα χρησιμοποιείται τα τελευταία τρία χρόνια έχει δημιουργήσει κάποια, ένα προηγούμενο σε ό,τι αφορά δηλαδή τους φορείς οι οποίοι λαμβάνουν αυτές τις πρωτοβουλίες, η Επιτροπή δηλαδή. Και ελπίζω πως αυτή ακριβώς η προηγούμενη εμπειρία δεν θα αποτελέσει κόλλημα για την περαιτέρω εφαρμογή της πρωτοβουλίας. Τώρα, ε, το τι μπορεί να γίνει. Ε, ένα εκατομμύριο υπογραφέ, ένα εκατομμύριο πολίτε για την πρωτοβουλία, νομίζω πω δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αυτό γράφεται, αναφέρεται ω τέτοιο δηλαδή ω όρο τη ε, συνθήκε. Δεν ξέρω αν θέλουμε τροποποίηση τη συνθήκη δεν ξέρω κατά πόσο και αν γίνει αυτό πράγματι θα βλάκει πάρα πολύ δική μας επιτροπή, από εκεί και μετά. Ε, κάτι που πρότεινα, το οποίο βέβαια δεν αναφέρεται εδώ στην νομοθετησία, αλλά το πρότεινα, είναι να εξεταστεί η εμπειρία των κρατών μελών ε, σε περίπτωση που υπάρχουν αντίστοιχα εργαλεία. Για παράδειγμα η Λετωνία έχει ένα ισοδύναμο ε, ε, σύστημα δηλαδή μια ε, πρωτοβουλία ε, πολιτών που ισχύει σε εθνικό επίπεδο και δεν νομίζω πω οι διοργανωτέ λοιπόν έχουν εξετάσει την εμπειρία που υπάρχει στα κράτη-μέλη με τέτοιου είδου πρωτοβουλίε πολιτών. Μετά, κάποιε άλλε σχέσει που έχω κάνει σε ό,τι αφορά του πόρου εάν θέλουμε πράγματι να έχουμε μια αναθεώρηση στο μέλλον τη πρωτοβουλίας των πολιτών, δεν νομίζω ότι πραγματικά ε, δεν θα υπάρξουν, δεν θα υπάρξει αντίκτυπο στον κοινωνικό προπολογισμό. Όχι, θα υπάρξει, ε, θα επιβαρυνθούμε περισσότερο και αυτό για να λειτουργούν καλύτερα οι πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τη δυνατότητα δημιουργία ενό help desk ενός δηλαδή μιας, ε, ενός γραφείου προσφοράς βοήθειας σε κάθε κράτος μέλος όπου θα είναι δυνατό οι πολίτες να απευθύνονται σε αυτό το helpdesk και να λένε ότι θα ήθελα να ξεκινήσω μια πρωτοβουλία πολιτών για το τάδι το δίνα ζήτημα και το helpdesk να πει ότι να λέει ότι όχι αυτό είναι μια κακή ιδέα αυτή η πρωτοβουλία γιατί δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια σειρά δηλαδή από πρωτοβουλίες πολιτών απέτυχαν ακριβώς για αυτό το λόγο επειδή δεν αφορούσαν αρμοδιότητα της Ένωσης. Επίσης θα μπορούσαν ε, να δίνονται καλύτερες εξηγήσει και το επιθυμούμε αυτό, καλύτερες εξηγήσει από την πλευρά της Επιτροπής. Ε, είπαμε ακριβώς και το ανέφερα και προηγουμένως ότι υπάρχει αυτή η απόκληση μεταξύ της νομικής και της πολιτικής ε, πτυχής δηλαδή ε, χρειάζεται η Επιτροπή να δίνει περισσότερες και πολιτικής φύσης εξηγήσει όχι μόνο νομικής φύσης τώρα το, η ελάχιστη ηλικία αναφέρθηκε 16 έτη στην Αυστρία θα μπορεί δηλαδή έχει νόημα κάποιο ε, με ηλικία 16 ετών να μπορεί να είναι πολιτών. Δεν έχω κάποια πολύ έτσι, κατηγορηματική άποψη από αυτού του ε, ζητήματο. Πάντω υπάρχουν τμήματα τη κοινωνία των πολιτών που πραγματικά ασκούν πιέσει για να ε, υπάρχει μια τέτοια εφαρμογή. Μετά, ε, υπάρχει και το ζήτημα που έχει ε, αναφερθεί και στην ακρόαση η προσωπική ευθύνη των διοργανωτών. Δεν χρειάζεται ενδεχομένω να τροποποιηθεί σε σχέση με αυτό το ζήτημα η συνθήκη, αλλά πραγματικά ε, είναι κάτι σημαντικό ότι συχνά δεν γνωρίζουν οι διοργανωτέ ποια είναι η προσωπική ευθύνη που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο μια πρωτοβουλία πολιτών. Για κάθε πρωτοβουλία που θα ξεκινάει θα πρέπει να γίνεται μια συζήτηση είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων υπό την εποπτεία, κάτι την άποψη, της δικής μας Επιτροπής και της Επιτροπής Αναφορών. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται και εκ των υστέρων μια συζήτηση. Νομίζω πως υπάρχει δηλαδή εδώ ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Δεν είναι δηλαδή γνωστό και υποψιάζομαι ε, ότι πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν περί τίνος ε, πρόκειται στις 24 ε, δηλαδή γλώσσες διαφορετικές και δηλαδή η κλασική αντίδραση είναι πρωτοβουλία πολιτών τι ακριβώς είναι αυτό, η πρώτη φορά τα ακούω Άρα λοιπόν ε, τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι εθνικές αντιπροσωπείες έχουν κάνει κάποια βήματα εδώ αλλά δεν έχουν κινηθεί αρκετά μακριά. Ε, υπάρχει και ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την καταχώρηση των υπογραφών. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ υπάρχουν 28 διαφορετικά συστήματα. Δηλαδή σε κάθε κράτος μέλους εφαρμόζεται ένα διαφορετικό σύστημα, ε, το είπα δηλαδή, ε, στην Ουγγαρία. Προτού για παράδειγμα μπορέσω να βάλω το δικό μου όνομα σε μια ε, πρωτοβουλία θα πρέπει να αναφέρω για παράδειγμα το όνομα γένους της μητέρας μου. Οι να γνωρίζουν για παράδειγμα κάποια άλλη, ένα άλλο σύστημα. Δεν ξέρω τέλος πάντων φτάνουμε σε ένα επίπεδο δηλαδή πραγματικά παραλογισμού ε, σε ό,τι αφορά την καταχώρηση μιας ε, υπογραφής. Ποια είναι δική μου ιδέα. Θα πρέπει να εξετάσουμε και την πτυχή της ψηφιακής ε, ιδιότητας του πολίτη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή δηλαδή ενδιαφέρεται για μια τέτοια προσέγγιση και εμένα μου αρέσει. Και από εκεί και μετά κάποιες από τις ε, τροποποίησεις που έχει ζητήσει η κοινωνία των πολιτών προϋποθέτουν τροποποίηση της συνθήκης και κατά συνέπεια εγώ λέω ότι σε σχέση με αυτές τις προτάσεις όχι δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν πρέπει να το κάνουμε. Και έχουμε την έκθεση ε, που ε, ανέφερα στην αρχή και εκδόθηκε 1η Απριλίου, είναι αρκετά σύντομη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε μια μεγάλη αναθεώρηση που θα είναι έτοιμη γύρω στο Δεκέμβριο. Ε, ελπίζω λοιπόν πως ε, οποιοδήποτε θα είναι το τελικό κείμενο της δικής μου νομοδότησης θα συμβάλλει σε αυτή την αναθεώρηση της Επιτροπής προκειμένου να βελτιωθεί ως εργαλείο. Πραγματικά θέλω πραγματικά να καταστεί ένα βιώσιμο, ένα αποτελεσματικό εργαλείο γιατί είναι μπορεί να καταστεί πολύ χρήσιμο ειδικότερο σε ό,τι αφορά ακριβώς την ε, δημιουργία ενός ισχυρότερου δεσμού μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σοσιαλιστές κύριε Κάουφμαν. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ε, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σόπφλιν για αυτό το ε, σχέδιο έκθεσης. Πραγματικά το διάβασα με μεγάλη μου χαρά. Περιλαμβάνει μια σειρά από ιδέες και τοποθετήσεις τις οποίες υποστηρίζω εμφαντικά και ε, είμαι πεπισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ε, Πολιτών μπορεί ε, να καταστεί περισσότερη φιλική προς τους πολίτες, ειδικότερα αν εφαρμόσουμε τις προτάσεις εδώ που περιλαμβάνει ο εισηγητής μας. Ο κύριος Σόφλιν μόλις τώρα ανέφερε πως η Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπέβαλε πρόσφατα και μία έκθεση η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική και για τις ε, διαβουλεύσεις που κάνουμε εμείς εδώ γιατί περιλαμβάνει μία σειρά από δεδομένα αλλά και εκτιμήσεις ως προς το τι λειτουργήσε καλά στον πλαίσιο των πρωτοβουλειών και τι όχι τόσο καλά οπότε θα πρέπει να διαβάσουμε πολύ προσεκτικά ε, την έκθεση αυτή αλλά και τη μελέτη που αναφέρθηκε μόλις τώρα στο πλαίσιο δηλαδή και τις ακροματικές διαδικασίες που είχαμε και η οποία ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σειρά από τα οποία υποστηρίζω πλήρω, αλλά θα ήθελα να τα θίξω εδώ και να κάνω κάποια σχόλια. Ε, τα σημεία τα οποία υποστηρίζω εμφατικά, λίγα να αναφέρω, ο κύριος Σόφριν το ανέφερε μόλις τώρα, δημιουργία δηλαδή γραφείων σε ό,τι αφορά την υποβολή πρωτοβουλίων πολιτών από την πλευρά της Ευρωπαϊκής ε, ε, Επιτροπής, δηλαδή μέσω ε, γραφείων επαφής με τους πολίτες. Μου φαίνεται πολύ σημαντική αυτή η πτυχή, ειδικότερα επειδή πολλοί διοργανωτές πρωτοβουλειών πολιτών μας είπαν επανειλημμένα ότι υπάρχει μεγάλη νομική αβεβαιότητα ως προς το τι ακριβώς περιλαμβάνεται στην ε, αρμοδιότητα, στο, στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής και τι όχι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνουν περισσότερη υποστήριξη οι διοργανωτές. Και νομίζω πως κατά συνέπεια η δημιουργία ε, τέτοιων γραφείων θα ήταν πολύ χρήσιμο. Ε, αναφέρομαι εδώ βέβαια στην παράγραφο 2. Ο κύριος Σόπλιον επίσης ανέφερε ότι σε περίπτωση απόρριψη μια πρωτοβουλία ε, πολιτών θα πρέπει πράγματι να παρέχει μια πολύ περιστατωμένη ε, αιτιολόγηση. Αυτό πράγματι καταδεικνύεται και από την εμπειρία που έχουμε συλλέξει κατά ε, τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή συχνά οι διοργανωτέ δεν γνώριζαν πώ ακριβώ να ερμηνεύσουν το κείμενο τη εξήγηση που ελάμβαναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή δεν ήταν αρκετή δηλαδή εξήγηση για να την καταλάβουν οι πολίτες. Άρα λοιπόν κάτι θα πρέπει να αλλάξει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, πολύ ενδιαφέρουσα ε, θεωρώ την πρόταση που κάνετε υπό την παράγραφο 5, ε, δηλαδή κατά την καταχώρηση ε, μίας πρωτοβουλίας πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο του να επιτρέψει να εγκρίνει ενδεχομένως τμηματικά μια πρωτοβουλία για παράδειγμα η πρωτοβουλία που αφορούσε τα δικαιώματα των μειονοτήτων ε, οδήγησε σε κάτι τέτοιο. Ήταν δηλαδή ιδιαίτερα εκτεταμένη και έχουμε βέβαια και την διαδικασία η οποία τρέχει ακόμα. Στην ακρόαση ακούσαμε και έναν εκπρόσωπο αυτής της πρωτοβουλίας. Σε κάθε περίπτωση εφόσον υπάρχει υπήρχε και για ε, την εν λόγω ε, πρωτοβουλία μια δυνατότητα αυτός ακριβώς τμήματικής έγκρισης ε, δεν θα οδηγούμασταν στο δικαστήριο αυτή τη στιγμή. Αναφέρεστε στο ζήτημα του λογισμικού υπό την παράγραφο 6, αναφέρεστε επίσης και στην χρηματοδοτική υποστήριξη για τις πρωτοβουλίες πολιτών. Έχουμε υποβάλει ούτως ή άλλως και υιοθετήσει για σχετικέ ε, τροπολογίε, ε, ε, τι οποίε θέσαμε στην Επιτροπή Προεπιλογισμών αλλά δυστυχώ δεν έγιναν δεκτέ από εκείνη σε κάθε περίπτωση στο πρόγραμμα Ευρώπη για του για, τους πολίτες είναι ένα καλό όργανο για την περαιτέρω χρηματοδότηση. Τώρα κάποια ερωτήματα. Αναφερθήκατε στην ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη υπό την παράγραφο 9. Κύριε Σόφλιν, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα, αλλά πότε θα προκύψει αυτή η ψηφιακή ηθαγένεια. Δηλαδή ενδεχομένως να χρειαστεί αρκετός ε, χρόνος εφόσον πράγματι τελικά δημιουργηθεί, συσταθεί ως τέτοια. Εκείνο όμως που εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι μια όσο το δυνατό ταχύτερη επανεξέταση του σχετικού κανονισμού και μια, ένα πιο πρακτικό αν θέλετε χαρακτήρα ε, των πρωτοβουλειών. Ε, και εδώ αναφερόμαστε και στους ε, αριθμούς ταυτοποίησης. Δηλαδή, ε, γνωρίζετε πως η κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή, σε διάφορα κράτη-μέλη προκειμένου να είναι δυνατό να πιστοποιηθεί η υπογραφή των πολιτών πρέπει να καταχωρούν εκεί μια, έναν αριθμό ταυτότητας, ένα ID number. Στη δική μου χώρα δεν χρειάζεται αυτό και οι διοργανωτές των πρωτοβουλίων πολιτών μας λένε ότι αποτελούν ε, ακριβώς αυτές οι αναφορές των αριθμών ε, ταυτοποίησης ένα μεγάλο εμπόδιο ε, στο πλαίσιο της υλοποίησης τέτοιων πρωτοβουλειών. Οπότε θα ήθελα εγώ να προσπαθήσουμε να εγκαταλείψουμε αυτή την ιδέα του αριθμού ταυτοποίησης στο πλαίσιο της πιστοποίησης δηλαδή των υπογραφών. Για το μέλλον δηλαδή θα ήταν κάτι τέτοιο πολύ ενδιαφέρον. Είδαμε και για παράδειγμα την ε, διαδικασία όπου η Σουηδία που έκανε μια πρόσφατη ε, για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις ε, μια πρόσφατη πρόφαση, πρόταση συγγνώμη, για να μην χρησιμοποιούνται τα ID numbers αντιθέτως η Μάλτα πρότεινε να χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από εκεί και μετά στην παράγραφο 10 αναφέρεστε σε ένα ζήτημα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε αλλά εδώ μας λέτε κύριε Σόφλιν ότι η ε, προσωπική ευθύνη θα πρέπει να είναι δυνατόν να επεκτείνεται σε ε, εθελοντικά συμμετέχοντες και υποστηρικτές της ε, λόγω πρωτοβουλίας. Μήπως μια τέτοια διατύπωση θα ήταν όμως αποθαρρυντική για άτομα τα οποία θέλουν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια πρωτοβουλία ίσως ε, καλή είναι η υπόλοιπη διατύπωση της ε, παραγράφου, δηλαδή στο τέλος της παραγράφου 10, όπου αναφέρουμε ότι θα πρέπει να είναι γνωστό ε, ποια είναι, σε ποιο βαθμό εκτείνεται η προσωπική ευθύνη, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά τώρα την προθεσμία για την επιβεβαίωση των υπογραφών, υπό την παραγράφο 11 δηλαδή, ε, εδώ ε, προτείνει ο κύριος Σόφλιν μια παράταση της σχετική προθεσμίας ε, κατά ένα έως δύο μήνες. Δεν είμαι βέβαια κατά πόσο πραγματικά είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα δηλαδή εδώ, εκεί το όπως αναφέρεται και πολύ σωστά στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι άλλο. Τα κράτη-μέλη αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την καταχώρηση των υπογραφών γιατί δεν γνωρίζουν κατά πόσο η πρωτοβουλία πολιτών τελικά θα εγκριθεί από την Επιτροπή αργότερα ή όχι. Δηλαδή, γιατί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με μια πρωτοβουλία χωρί να ξέρει εκ των προτεραιών αν υπάρχει πιθανότητα να εγκριθεί. Άρα λοιπόν εκεί ε, προκύπτει το πρόβλημα και όχι στο πλαίσιο τη ίδια δικασία τη καταχώρηση των υπογραφών. Κατά συνέπεια δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να παραταθεί η σχετική προθεσμία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σοδευτική προθεσμία. Ε, κάνετε μια σχετική αναφορά στην ε, παράγραφο 11 και στο παράγραφο 7 κάνετε και μια αναφορά. Ουσιαστικά δηλαδή ε, με αυτές τις δύο αναφορές ε, μας προτείνετε δύο διαφορετικές λύσεις. Οπότε εγώ θα ήθελα να ταχθώ κατηγορηματικά περί της μίας από αυτές τις λύσεις. Ε, μας λέτε δηλαδή ε, υπό την παράγραφο 11 η σχετική προθεσμία θα πρέπει να πάει στους 18 αντί για τους 12 μήνες. Κατά τη δική μου άποψη, ε, μια προθεσμία 18 μηνών για τη συγκέντρωση των υπογραφών, ειδικά στην περίοδο που πραγματικά αλλάζει γρήγορα η νομοθεσία, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ ρεαλιστικό. Ε, ίσως θα πρέπει να υπάρχει μια αυτοματοποίηση ό,τι αφορά την καταχώρηση ε, μια ε, πρωτοβουλία και από την άλλη συγκέντρωση των σχετικών υπογραφών. Αυτό είναι ακριβώ και το ειδικότερο διοικητικό, αν θέλετε, διαχειριστικό πρόβλημα για του διοργανωτέ. Δηλαδή, όταν θα γνωρίζει ένα διοργανωτή ότι ε, από τη στιγμή που ξεκινάμε τη συγκέντρωση, από τότε αρχίζει να τρέχει και η προθεσμία των 12 μηνών, τότε μπορούν να, ξέρουν, να οργανωθούν καλύτερα. Γνωρίζουν δηλαδή ότι έχει καταχωρηθεί η πρωτοβουλία και γνωρίζουν ότι για τους συγκεκριμένους 12 μήνες εκείνο που πρέπει να κάνουν είναι να συγκεντρώσουν τις υπογραφές. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν το σκεπτικό ότι πραγματικά να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία και περισσότερη, αν θέλετε, ε, ε, ε, πιο δραστήρια συμμετοχή στη συγκέντρωση των υπογραφών, αλλά θα πρέπει να, να, να βρεθεί διαφορετικά η λύση και όχι με την παράταση της προθεσμίας. Επίσης έχω ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά την διατύπωση παραγράφου 13. Το διάβασα αυτό το κείμενο εδώ και στα αγγλικά και στα γερμανικά. Δεν είμαι σίγουρο αν καταλαβαίνω σε τι ακριβώς αναφέρεστε, λέτε ότι θα πρέπει η Επιτροπή να ξεκινήσει ε, μια, της προετοιμασία νομικής πράξης ε, εντός 12 μηνών μετά, δηλαδή από την έγκριση μιας ε, πρωτοβουλίας ε, πολιτών. Μας λέτε δηλαδή ότι τι, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδρά νομοθετικά εφόσον έχει εγκρίνει μια πρωτοβουλία πολιτών. 12 μήνες λοιπόν λέτε για την προετοιμασία μιας αντίδρασης. Δηλαδή η αντίδραση τι μπορεί να είναι. Ότι ε, του χρόνου θα εκδοθεί μια λευκή βίβλος από εκεί και μετά θα υπάρχει ακροαματική διαδικασία και οτιδήποτε άλλο. Άρα δηλαδή μπορεί να ε, γίνει πάρα πολύ ε, χρονοβόρα μια τέτοια διαδικασία. Οπότε θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο καλύτερα τι ακριβώς εννοείται στην παραγραφό 13. Ε, τέλος, για να κλείσω ε, κυρία Πρόεδρε, ε, μας είπατε ε, κύριε Σόπφλιν ότι ε, το ζήτημα της ελάχιστη ηλικία δεν είναι πολύ σημαντικό για σας, αλλά κατά τη δική μου άποψη είναι εξαιρετικά σημαντικό. αυτό άκουσα εγώ. Α, είστε ουδέτερο, είπατε. Ναι, είναι καλύτερα που μας λέτε ότι είστε ουδέτερο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το συζητήσουμε μεταξύ μα. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε με μία νομική πράξη, δηλαδή ε, πιο, ε, όχι τόσο σημαντική αν θέλετε, δηλαδή πραγματικά έχουμε κάποιους ε, ε, ε, πολίτε οι οποίοι με την υπογραφή τους αποφασίζουν αν θέλουν να συμβεί κάτι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο αναλυτοί μπορούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή το ότι δίνεται αυτή η δυνατότητα στους 16χρονους στην Αυστρία δεν ξέρω κατά πόσο είναι ενδεδειγμένο. Στο υπόλοιπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ως ελάχιστη ηλικία τα 18 έτη. Ε, νομίζω πως θα πρέπει δηλαδή να προσπαθήσουμε από την πλευρά μας να επιβληθεί μια ενιαία, ε, ένα ενιαίο όριο ηλικίας. Δηλαδή για να ξέρουμε κατά πόσο ε, θα θεωρούμε ότι ένα, ένας πολίτης είναι σε θέση να ταχθεί όχι υπέρ μιας ιδέας στο πλαίσιο της Ευρώπης. Οπότε νομίζω πως ένας 16χρονος δεν είναι σε θέση να το πράξει αυτό. Ε, πάντως εν γέννη θεωρούμε πως πραγματικά έχουμε να κάνουμε ένα εξαιρετικό σχέδιο ε, έκθεσης και νομίζω πως θα πρέπει να αναφέρεται ρητά εν λόγο κείμενο ότι χρειαζόμαστε και να εκτιμάμε του, του σχετικού κανονισμού, δηλαδή αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού, τόσο ώστε πραγματικά να μπορέσει να αναπτύξει το πλήρε δυναμικό τη και να αξιοποιήσει το πλήρε δυναμικό τη η πρωτοβουλία πολιτών και να αξιοποιείται στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό από του πολίτε. Και βέβαια εδώ και ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκφραστούν γιατί αν θέλουμε να τροποποιήσουμε τον κανονισμό και οι δύο νομοθέτες βέβαια θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαντόφσκι. Κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Σεπφλίν για το σχέδιο κειμένου. Είναι σαφές, εναργές, θέλει να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και τη σχετική πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και συμφωνώ με τις απόψεις του κειμένου. Για την νομοθεσία, το πιο σημαντικό είναι να υιοθετούμε νόμους οι οποίοι να μπορούν να εφαρμοστούν, ειδικά όταν αφορούν, αφορούν τους πολίτες. Επομένως, υποστηρίζω την πρότασή σας, η οποία θέλει να παρακάμψει τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Επίσης, συμφωνώ με την επέκταση της προθεσμίας για τη συλλογή υπογραφών και όπως και οι προλαλήσαντες, ο προλαλήσας μάλλον, να τονίσω ότι παράγραφος 13 είναι η πιο βασική παράγραφος. Έχει νόημα να εισάγουμε τις σωστές αλλαγές, τις σωστές αλλαγές στην νομοθεσία. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να δρά κατά το δοκούν. Εγώ λοιπόν ερμηνεύω την παράγραφο με καλή θέληση ως μια υπόσχεση ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία που πληρεί κάποια κριτήρια και υποστηρίζεται από τον επαρκή αριθμό πολιτών να γίνει μια νομοθετική πρόταση. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την παράγραφο 13, θα μπορούσαμε να κάνουμε και διευκρινήσεις. Αλλά νομίζω ότι η παράθυρα αυτή είναι βασική για να προχωρήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να δρά όπως θέλει γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να το κάνει, μπορεί να απορρίψει και προτάσεις που πληρούν ακόμα όλα τα τυπικά κριτήρια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά την προσοχή στο σημείο 13 και ευχαριστώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που εντοπίσατε τα βασικά στοιχεία ούτως ώστε το κείμενο αυτό να είναι, το μέσο αυτό να είναι πραγματικά αποτελεσματικό. Μας Θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο ενεργητικοί για να προωθήσουμε μια τέτοια πρωτοβουλία. Ξέρετε ποιες δυσκολίες υπάρχουν σε αυτή την πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή. Και επιπλέον υπάρχει και το πρόβλημα της αφαίρετης δράσης της Κομισιόν. Εάν απογοητεύσουμε τους ε, πολίτες που είναι πιο δραστήριοι και ενεργητικοί, νομίζω ότι θα κάνουμε τεράστια ζημιά. Πιο μεγάλη ζημιά θα κάνουμε, παρακαλώ. Θα πρέπει λοιπόν ε, να εντοπίσουμε τα προβλήματα και νομίζω το, το κάνετε πολύ καλά κύριε Σιγητά. Το θέμα της ανάλυσης που περιμένουμε για όλους τους λόγους για τους οποίους αποτυγχάνουν αυτές οι πρωτοβουλίες όλα αυτά τα στοιχεία που εντοπίζει η έκθεση. Και βεβαίως πρέπει να κάνουμε μια δουλειά μαζί με την Επιτροπή Αναφορών. Αλλά το θέμα του Μητρώου του, των υπογραφών, το θέμα ότι δεν μπορούμε να έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα νέα εργαλεία που έχουμε, τα ψηφιακά, τα μη αναλογικά δηλαδή, για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτά τα θέματα όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, όλα αυτά που είπε η κυρία Κάφμαν, όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, ούτως ώστε να προτείνουμε αυτά που πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο από την πλευρά του, τόσο ώστε να βοηθήσει την Κομισιόν να δρά και πιο υπεύθυνα. Ε, δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που στο παρελθόν αντιμετώπισαν δυσκολίες ε, λόγω ερμηνείας, λόγω μητρώου, λόγω ασυνέπειας σε ό,τι αφορά τους κανόνες εφαρμογή, εφαρμογής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σοβαροί ε, και νομίζω ότι ξεκινήσατε μια δουλειά αξιοσημείωτη και σας συγχαίρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Μπάρμπαρα Σπινέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Σέπφλιν για το πλαίσιο παρουσίασης της κατάστασης, για τα, τις εκκλήσεις που κάνει, για την ψηφιακή ηθαγένεια κυρίως, για την απλούστευση των διαδικασιών συλλογής υπογραφών. Υπάρχει ένα σημείο, το οποίο νομίζω είναι σημαντικό, το οποίο θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε περισσότερο στο σημείο 13 για την συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί για το follow-up. Η πρωτοβουλία των πολιτών περνά από βαθύτατη κρίση. Γιατί δεν είναι σαφές αν υπάρχει ασφάλεια για τους πολίτες ότι θα δοθεί συνέχεια στα αιτήματά τους. Γι' αυτό λοιπόν διερωτώ με δύο πράγματα. Πρώτον, όταν ζητάμε από την Κομισιόν να εκπονήσει μία νομοθετική πράξη. Μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία αποδοχής με επιτυχής ΕΠΠΠ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την πρωτοβουλία των πολιτών που συγκεντρώνει ας πούμε τα εκατομμύρια πολιτών που απαιτούνται. Μία πρωτοβουλία που γίνεται αποδεκτή αλλά δεν υπάρχει μια, καμία συνέχεια. Δεν υπάρχει κανένα follow-up παρόλα αυτά. Παραδείγματο χάρη τη πρωτοβουλία για το νερό. Έγινε κάτι τέτοιο, όπου δεν υπήρξε κανένα follow-up. Και το δικαίωμα των πολιτών, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν ακριβώ αυτή η πρωτοβουλία για το νερό, εν πάση περιπτώσει. με αν είναι χρήσιμο λοιπόν να έχουμε μια εναλλακτική φόρμουλα για πρωτοβουλίες πολιτών που συγκεντρώνουν τον αριθμό υπογραφών, αλλά δεν γίνονται αποδεκτές από την Επιτροπή. Τι γίνεται με τις πρωτοβουλίες που τις κάνει δεκτές η Κομισιόν, αλλά που δεν υπάρχει παρόλα αυτά κανένα follow-up, καμία συνέχεια δεν δίνεται. Αυτά είναι, δύο, είναι διαφορετικές περιπτώσεις που θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Ο κύριος Θερικάμπρας έχει φύγει, δεν θέλει να μιλήσει. Ο κύριος Φάμπιο Μάσιμου είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Σέπλιν, για τη δουλειά που έκανε, διαβάζοντας την έκθεση συνειδητοποίησα την πολύ προσεκτική δουλειά που έκανε, τις ιδέες που είχε, τις συγκεκριμένες προτάσεις. Έκανε δηλαδή μια έρευνα πολύ σημαντική για το τι έχει γίνει με τις διάφορες πρωτοβουλίες. Τα διάφορα πήρε feedback δηλαδή από όλα όσα έχουν γίνει. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το 6, 9, το 6, 7, 8, 9 και 11. Ε, αυτοί που συμμετείχαν σε επιτροπές αλλά και συμμετείχαν σε πρωτοβουλίε, είπαν ότι ένα βασικό πρόβλημα ήταν ότι είναι πάρα πολύ επαχθή η όλη διαδικασία και οικονομικά. Οποιοδήποτε αποφασίζει να κάνει αυτό το, αυτή την προσπάθεια για άσκηση άμεση δημοκρατία προσκούει σε πολλά εμπόδια, πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να προσκούρουμε στο πρόσκομα ενός πολύ σημαντικού οικονομικού άχθους. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ε, αυτό το θέμα και να απλουστεύσουμε ε, τον τρόπο συλλογής υποψηφιακά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και να μειώσουμε το κόστος και να απλουστεύσουμε τη διαδικασία. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι σε ό,τι αφορά το σημείο 13, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε και η κυρία Σπινέλη προηγουμένως, μην ξεχνάμε, το εξή. Υπόθηκε προηγουμένω. Υπάρχει μια αποσύνδεση σαφέστατη ανάμεσα στον πολίτη, τον Ευρωπαίο πολίτη και στην ταυτότητά, την ευρωπαϊκή του ταυτότητα. Ήταν ένα από τα σημεία που έχουν αναφερθεί. Συμφωνώ με αυτό. Συχνά αυτά τα εργαλεία δεν είναι αρκετά γνωστά, δεν είναι ε, ευρέως γνωστά. Και έχω την αίσθηση ότι μετά από τόση προσπάθεια φτάνουμε σε αποτελέσματα που δεν είναι αναλογικά με όλη την προσπάθεια που έχουμε καταβάλει. Δηλαδή συχνά υπάρχουν αυτά τα πράγματα, αλλά δεν δίνεται καμία συνέχεια. Δεν αξιοποιούνται. Νομίζω ότι θα πρέπει να, αξιοποιήσουμε, να ζητήσουμε από την Κομισιόν ε, για κάθε πρωτοβουλία η οποία συγκεντρώνει όλα τα τυπικά προσόντα να δοθεί συνέχεια. Γιατί αλλιώς ας πούμε, ακυρώνουμε την ε, πρόθεση των πολιτών, την, την επιθυμία των πολιτών. Και παρότι, ας πούμε, Υπάρχει ε, ενδιαφέρον, πούμε, από πολίτες, πολλούς πολίτες, ε, βλέπουν οι πολίτες ότι δεν δίνεται καμία συγκεκριμένη συνέχεια. Πέφτει στο κενό ε, η προσπάθειά τους. Όταν θα μπούμε και στις τροπολογίες θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να υπάρξει ένας καλός ορισμός προς αυτήν την κατεύθυνση αυτών των στοιχείων που σας είπα και ελπίζω να υπάρξει μια πλατιά συμφωνία όλων των μελών της Κομισιόν γύρω από αυτό ακριβώς το σημείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το εργαλείο και διαπαιδαγωγικό. Αν έχουμε ένα εργαλείο που λειτουργεί καλά, έτσι, εάν του δώσουμε ας πούμε, φωνή στο, στη διαδικασία λήψη των αποφάσεων, ίσως τότε, μετά από κάποια χρόνια, εντάξει, ίσως είναι πρόημο αυτό που θα σας πω, αλλά μου αρέσει να ονειρεύομαι, και καλό θα ήταν να γίνουν ενδεχομένως και ευρωπαϊκά ρεφερέντουμ ε, ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα. Εντάξει, είναι ένα όνειρο σας είπα, αλλά γιατί όχι. Ε, μπορεί να είναι η απαρχή ενό πράγματος πολύ πιο ισχυρού, πολύ πιο έντονου. Ευχαριστώ. Η, κυρία Κάρμεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very much, Madam Chairman. Κυρία Πρόεδρε, έχω μερικά γενικά σχόλια και έχω και κάποιες απαντήσεις να δώσω σε θέματα που εθίγησαν κατά τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις συζητήσεις στις άλλες επιτροπές. Μια συζήτηση αναβλήθηκε σήμερα αλλά θα γίνει το Μάιο και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο καταλείπει αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας διότι είχαμε πολιτικό υλικό αλλά ε, δεν ήταν θεσμικά σε θέση να προχωρήσει. Τώρα έχουμε μια μεγάλη και λεπτομερή ανάλυση, της ε, ανάλυση, του θέματος. Ε, Βεβαίω όλα αυτά δεν είναι η πολιτική θέση του θεσμού. Συνεπώς το ψήφισμα το οποίο ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει μετά τους θερινές διακοπές θα συμπληρώσει τη θέση του την ευρύτερη και ελπίζουμε ότι και το Συμβούλιο θα αρχίσει να συζητά την έκθεσή μας για να το γυρθεί σε συμπεράσματα. Δηλαδή μέσα στη χρονιά θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εικόνα και να καταλάβουμε και καλύτερα την κατάσταση. Στην έκθεσή μας λέμε με σαφήνεια ότι ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς θεωρεί ότι ο μηχανισμός μετά από δύο χρόνια, δηλαδή ο μηχανισμός της πρωτοβουλίας των πολιτών εφαρμόζεται ικανοποιητικά. Βεβαίως υπάρχουν λήψεις, τις αναφέρουμε δε ε, με σαφήνεια στην έκθεσή μας χωρίς να τοποθετούμεθα για την επόμενη προσέγγιση αλλά όλα αυτά ε, είναι μια έκθεση προς τους ενδιαφερόμενους όπως εσείς και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ενδεχόμενες μεταβολές αργότερα μέσα στη χρονιά μπορεί να καταλήξουμε ότι πρέπει να μεταβληθούν οι κανόνες. Ευχαρίστως τότε θα διερευνήσουμε τις δυνατότητες. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν προσεκτικά. Σπάνια ο κανονισμός αναθεωρείται μετά από τρία χρόνια. Είναι νωρί λοιπόν, δεν θέλουμε να προτρέξουμε ανοίγοντας μια νομοθετική αναθεώρηση συνεπάγεται κινδύνους και αυτό Βεβαίως ευχαρίστως να εξετάσουμε τις ελλείψεις. Η έκθεσή σας, το σχέδιο της έκθεσής σας ε, θέτει λίγο πολύ τα ίδια θέματα που θέτουμε και εμείς στην έκθεσή μας. Έχουμε και την έρευνα του Ombudsman, δικιά του έρευνα, Δηλαδή έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και γενικά συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την έκθεση και τις συζητήσεις. Ένα πράγμα είναι σημαντικό, να ξεχωρίσουμε και να μην ανακατέψουμε ώστε το κοινό να καταλαβαίνει, να ξεχωρίσουμε λέω τις μεταβολές που μπορούν να γίνουν μέσα στο πλαίσιο του σημερινού νομικού πλαισίου και των μέτρων που συνεπάγονται μεταρρύθμιση του ισχύοντος πλαισίου. Υπάρχουν δηλαδή ε, σημεία τα οποία ε, συνεπάγονται μεταβολή του σημερινού κανονισμού, όπως η επιμήκυνθηση. Αλλά είναι σημαντικό ταυτόχρονα να πούμε ότι υπάρχουν και θέματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν απλά βάσει του τρέχοντος πλαισίου όπως οι απαιτήσει ε, των βασικών στοιχείων. Ε, δεν είναι κάτι που συζητήσαμε σήμερα, αλλά σαφέστατα αποκλείει μεγάλο αριθμό πολιτών από τη προσφυγή σε αυτή την πρωτοβουλία. 1η Μαρτίου η Κομισιόν υιοθέτησε μια άλλη καταπαραχώρηση, κατεξουσιοδότηση πράξη, καλώντας τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μια πιο επικοδομητική προσέγγιση και απλούστερους κανόνες ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να χρησιμοποιούν αυτόν τον μηχανισμό. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, ότι με το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση σημερινή μέσω των κατεξουσιοδότηση πράξεων της Κομισιόν. Έχουμε λοιπόν ανοίξει και το νέο λογισμικό, το οποίο είναι μια βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο. Έχουμε διασύνδεση με τα κοινωνικά μέσα, δηλαδή αν θέλετε και από την άποψη του λογισμικού έχουμε βελτιώσει τα πράγματα. Τώρα, ως προς την πολιτική συζήτηση στην οποία αναφέρεται ο εισηγητής, έχουμε τις ακροάσεις, μια ακρόαση θα γίνει στην Επιτροπή Άγκρη, σύντομα και είναι, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία της ακρόασης για να έχουμε μια πραγματική πολιτική συζήτηση και να ακούσουμε διαφορετικές απόψεις ώστε να συμμετάσχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι και όχι μόνο οι οργανωτές. Έχουμε λοιπόν μόνο Τρεις μήνες για να ανταποκριθούμε στην πρωτοβουλία των πολιτών είναι πολύ σύντομα για να κάνουμε μια δημόσια διαβούλευση. Συνεπώς η ακρόαση στο Κοινοβούλιο είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για μια ευρύτερη συζήτηση και την εμπλοκή περισσότερων ενδιαφερομένων. Ακόμη θα ήθελα να αναφερθώ και στις μεταφράσεις, τις οποίες αναφέρομαι και στην έκθεσή, μας με ρεαλισμό και καλή θέληση. Υπήρξε συμφωνία ότι η Κοινωνική Επιτροπή θα προσφέρει τις υπηρεσίες ε, μεταφράσεων και αυτό δείχνει πώς μπορούμε να πετύχουμε βελτιώσεις μέσα στο σημερινό πλαίσιο, όπως σας έλεγα στην αρχή. Ακόμη κάποια θέματα. Το Help Desk, το Europe Direct είναι ένα κέντρο εξυπηρέτηση. Ε, που μπορεί να βοηθήσει την ενίσχυση των γνώσεων των πολιτών. Υπάρχει πο, πολύ λίγοι οργανωμένοι χρησιμοποιούν αυτούς τους μηχανισμούς. Απορρίφθησε η χρησιμοποίηση αυτού του ενδεχόμενου σε κάποιο βαθμό ε, πρέπει να εξηγήσουμε σωστά τις αρνήσεις αυτές ε, εκ μέρου μας και δίνουμε τις επεξηγήσεις στο διαδίκτυο. Υπήρξαν δηλαδή πρωτοβουλίες οι οποίες μετά την ανάλυση των επιχειρημάτων μας ξαναδιατύπωσαν την πρότασή τους και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή διαβάζοντας και τις επεξηγήσεις μας μπορεί κανείς να βγάλει και κατάλληλα συμπεράσματα. Όσον αφορά την εγγραφή ή την μερική εγγραφή γενικά, το δικαστήριο θα μας δώσει κατευθύνσεις πάνω σε αυτό. Ελπίζουμε ότι δεν θα καθυστερήσουν ε, την απόφαση και έτσι θα υποφεληθούμε από την άποψή τους. Όσον αφορά την επέκταση, την παράταση της περίοδου, πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα η πρωτοβουλία δεν έχει πετύχει ένα εκατομμύριο υπογραφές, όχι μόνο δε για την προθεσμία των 12 μηνών και για άλλους λόγους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τζόρτς τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και την Κομισιόν, την κυρία Πράιζεν. Ε, ευχαριστώ για τις τροπολογίες σας θα συζητήσουμε την σχετική ημερομηνία. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα την ερώτηση κόφρα σε σχέση με την παράγραφο 13. Στο αγγλικό λέει παροτρύνει την Κομισιόν να συντάξει μια νομοθετική πράξη μέσα σε 12 μήνες από την αποδοχή. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές και προχωρά περισσότερο αν θέλετε από τον υφιστάμενο κανονισμό. Τουλάχιστον αυτό είχα κατά νου. Ε, δηλαδή δίνουμε μία συνέχεια που απαιτείται. Νομίζω συμφωνείτε όλοι σε αυτό. Τώρα υπήρχε και κάτι άλλο που ήθελα να πω για να κοιτάξω τις σημειώσεις μου. Η κυρία Πράιζινγκ αναφέρθηκε στους πολίτες που ζουν σε χώρες εκτός της δικιάς τους είναι πολύ δύσκολο να υπογράψουν πρωτοβουλίες και αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Δεν ξέρω ακριβώς πώς πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να το σκεφτούμε. Ακόμη, υπάρχει ένα άλλο σημείο που ίσως δεν το έχω αποσαφηνίσει αρκετά. Όταν γίνεται μια κοινοβουλευτική ακρόαση, δεν θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στην Επιτροπή που θα επηρεαστεί από τη σχετική ακρόαση. Πρέπει να έχει ε, συμβολή από πολλές επιτροπές. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας για την συμβολή σας. Θα περιμένω τις τροπολογίες σας συγκεκριμένα και ελπίζω αυτός ο μηχανισμός να γίνει αποτελεσματικός. Ευχαριστώ, George. να πούμε ότι, ότι α, ε, 20 Μαΐου λοιπόν προτείνω όσο ε, προθεσμία για τον πολύ τροπολογιών, ένα μήνα από τώρα. Και μετά θα έχουμε ψηφοφορία στην Επιτροπή το Σεπτέμβριο πλέον. Δεν ξέρω τώρα κατά πώς δικαιολογείται να είναι ψηφοφορία το Σεπτέμβριο. Καλώς, περνάμε λοιπόν στο τελευταίο σημείο της σήμερας διάταξης, Ραμόν Χαουρέγγι, νομοδότηση σε ό,τι αφορά την κατάσταση ε, των θεμελιωδιών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μια γνωμοδότηση λοιπόν από την δική μας πλευρά προς την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Λόγω στον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, πρόκειται για μια γνωμοδότηση, για μια έκθεση από το 1993 η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ξεκινάει για να εξετάσει την κατάσταση. Ποια κατάσταση, το κατά πόσον δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να σας κάνω είναι ότι η έκθεση της ΛΥΜΠΕ είναι όχι τόσο εκτεταμένη όσο αυτή που λαμβάναμε τα περασμένα χρόνια. Νομίζω ότι επίτηδες το κάνουν. Θέλω να κάνουν μια γενικότερη αναφορά στην κατάσταση του κατά πόσο γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν αρκετές διαφορές σε σχέση πράγματο χάρη με την περασμένη έκθεση που μα έχει υποβάλει Λίμπε εκ μέρου του Λουί Μισελ. Είναι πολύ πιο λακωνική, είναι πολύ πιο ευσύνοπτη. Ωστόσο, αναγκαστικά απεικονίζει την κατάσταση στην Ευρώπη. Από πολλές απόψεις σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Γιατί η Ευρώπη ήταν πάντα ένας φάρος ε, πολιτισμού σε ό,τι αφορά την προάσπιση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η έκθεση θέλει να είναι γενικόλογη και κάπως αφηρημένη ως σε ό,τι αφορά τα συμβάντα που συνέβησαν αυτή τη χρονιά στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, τελικά δεν έχει αρκετά αναλυτική δύναμη, ε, δεν παρουσιάζει αρκετά έντονα τα όσα συμβαίνουν. Η έκθεση ε, για αυτή την έκθεση εμείς εκδίδουμε μία γνωμοδότηση εδώ στην ΑΦΚΟ. Η Επιτροπή Γυναικών, η ΠΕΤΗ και άλλη μία ε, εκπονούν γνωμοδοτήσεις προς τη ΛΥΜΠΕ. Έχουμε 7 μεγάλα τμήματα σε αυτήν. Καταρχάς τα θεσμικά, δηλαδή ε, ασφάλεια και ελευθερία, τα προβλήματα ισότητας, τα προβλήματα με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα θέματα αλληλεγγύης, και το κατά πόσον υπάρχει αλληλεγγύη λόγω της ε, ε λιτότητας, το θέμα της ε, εγκληματικότητας και της διαφθοράς και κατάσταση ε, των κρατήσεων σε κρατητήρια και σε φυλακές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σύντομα να σας πω ότι αυτή η έκθεση που παρουσίασε η ΛΥΜΠΕ έχει δύο βασικά στοιχεία που, ξεχωρίζουν, που πρέπει να τα προσέξουμε κατά την απόψή μου ιδιαίτερος. Από τη μία, αναφέρει την ιδέα ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι επιθυμεί να δημιουργηθεί μια στρατηγική, εσωτερική στρατηγική όπως ονομάζεται, μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επαγρυπνεί για τις πρακτικές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα θέματα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και υπάρχει και μια διαδικασία ε, εποπτείας ε, για το κατά πόσο γίνονται σεβαστές αυτές οι αρχές και ενσωματώνονται σε όλες τις νομοθεσίες. Και μια διαδικασία που ε, εποπτεύουμε τα κράτη-μέλη για το κατά πόσο υπάρχουν παραβιάσεις από μέρους τους. Αυτό υπάρχει στη συνθήκη, στις συνθήκες μάλλον, άρθρο 7. Όμως Υπάρχουν πολλέ προποθέσει ούτω ώστε η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο κτλ. να εγκαλέσει ένα κράτο μέλο γιατί παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το άρθρο 7 το προβλέπει αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δημιούργησε αυτή τη διαδικασία ούτω ώστε να υπάρχει μια πρακτική ας πούμε επιτήρησης, παρέμβασης αν θέλετε των θεσμικών οργάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κομισιόν και Συμβουλίου έναντι ενός κράτους μέλους. Όπως ε, λέει και το άρθρο 7 της συνθήκης, ε, πρέπει να υπάρχει μία μεγάλη πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 4 πέμπτα, έτσι, για να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Ε, η έκθεση λέει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα απέναντι σε αυτή τη διαδικασία που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, εγώ έχω έξι σημεία στη δική μου έκθεση, το, στο κείμενο που έχετε, και ελπίζω επ' αυτού να τοποθετηθείτε. Και πρόεδρε, μέχρι τις 21 του μηνός, 21 Απριλίου, έχουμε προθεσμία για σχόλια δικά σας. Λοιπόν, Το κείμενο αυτό είναι λίγο πιο μακροσκελέ από ό,τι συνηθίζεται σε γνωμοδοτήσει επιτρόπων όπω η δική μας. Σας παραπέμπω τώρα στο περιεχόμενο της εκθεσή μου, της γνωμοδότησής μου μάλλον, του κειμένου μου. Και μιλάω για την ανάγκη να επιμείνουμε περισσότερο στο, ε, νούμερο ένα στο ψηφίσμα νούμερο 1 της ΛΥΜΠΕ, όπου πρέπει να, όπου μιλάμε για το σεβασμό και την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Να κάνω και μια πολιτική αναφορά εδώ, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι τα συμβάντα τα οποία λαμβάνουν χώρα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας αναγκάζουν να κάνουμε ένα προβληματισμό ε, για να δούμε σε ποιο βαθμό έχουμε προχωρήσει ε, για να σεβαστούμε εντό αγωγικών τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελευθερία έκφρασης, ε, ε, δημοκρατικά δικαιώματα, διαφάνεια, ε, όλες τι προσδοκίες, εν που δημιούργησαν τα κράτη δικαίου μα. Η κατανομή των ρόλων ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία, νομοθετική εξουσία κτλ. και δικαστική εξουσία, το ισχύει στον πολιτών, και εν πάση περιπτώσει η, στάση του πολίτη απέναντι στο κράτος. Νομίζω ότι αυτή η θέση αποδυναμώνεται. Ε, πέρα από αυτό που προβλέπει το, το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Συμβόλαιο. Υπάρχουν διάφορα θέματα, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα, διάφορα ε, δικαιώματα τα οποία η κρίση τα υπέσκαψε. Είναι σημαντικό η Επιτροπή ΑΦΚΟ να κάνει ένα πρώτο προβληματισμό στην ανάγκη να επαναδιεκδικήσουμε την ουσία αυτών των δικαιωμάτων. Ε, υποτίθεται ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι η εμπροστοφυλακή ε, του μηχανισμού που προστατεύει αυτά τα δικαιώματα. Η ΑΦΚΟ επίσης είναι σημαντικό να κάνει και ένα προβληματισμό για το ατελεύτητο θέμα της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Ε, το κάνει η ΛΥΜΠΕ, αλλά η ΑΦΚΟ είναι επιτροπή κλειδί σε αυτό το θέμα και πρέπει να ζητήσει από την ε, Κομισιόν και, το Συμβούλιο την, ε, την επανεκκίνηση της διαπραγμάτευσης με το δικαστήριο, ούτως ώστε να υπάρξει προσχώρηση στη σύμβαση. μετά την απόφαση που έκανε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, που φρέναρε την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την έκθεσή μας είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή η διαπραγμάτευση πρέπει να προχωρήσει και να ε, τελεσφορήσει. Ε, η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Επίσης, ε, το κοινωνικό και εργατικό πλαίσιο ε, έχει υποβαθμιστεί. Είναι σημαντικό να το διεκδικήσουμε ξανά, όπως σας είπα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή, Χάρτα, ε, Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα είναι σημείο αναφορά για την προάσπιση αυτών των καθολικών δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων που σας έλεγα προηγουμένως. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Χάρτα δεν απεικονίζεται επαρκώ ε, στα κείμενά μα. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαρκώ στα κείμενά μα. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό κείμενο και εμπνέει, ε, και από αυτό εμπνέεται αυτό το ε, κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο χαρακτηρίζει την Ευρώπη τα τελευταία 50 χρόνια. Επίσης, υπάρχει ανάγκη να λάβουμε υπόψη μας ότι Κατά πάσα πιθανότητα το μεγάλο πρόβλημα που ανταμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ε, η μεταχείριση των ε, μειονοτήτων. Σωστά ε, λέγεται ότι η δημοκρατία είναι σεβασμός των μειονοτήτων. Δεν είναι τόσο το πώς λειτουργούν οι πλειοψηφίες. Το βασικό είναι οι πλειοψηφίες να σέβονται τις μειοψηφίες ή μειονότητες, ας πούμε. Εκεί φαίνεται η δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωσή μα έχει πάρα πολλέ μειονότητε και μειοψηφίε γενικά και δεν γίνονται πάντα σεβαστέ. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν αυτή την ιδέα, να... Ε, το να μπορεί η πολιτική και η εσωτερική στρατηγική που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Προστασία των Θεμελιωδών ομάδων θα πρέπει να έχει ως βασική εστίαση το γεγονό ότι υπάρχουν πάρα πολλέ μειονότητε. Δεν έχει νόημα να τι αναφέρω. Ε, τι έχετε στο μυαλό σα. Ε, ξέρετε πολύ καλά τα όσα συμβαίνουν, ε, τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω φύλου, λόγω ε, εθνοτικής προέλευσης, ε, λόγω σοξιολικού προσανατολισμού, θρησκείας κτλ. Θα πρέπει να συνεχίσει η Ευρώπη να είναι αυτός ο εκπολιτιστικός φάρος. Επειδή σέβεται τα δικαιώματα, επειδή προασπίζεται τα δικαιώματα ε, των ε, μειονοτήτων στην κοινωνική της πραγματικότητα. Γι' αυτό πρέπει να το πούμε αυτό. Και τέλος, υπάρχουν και τρεις σημαντικές πτυχές που είναι σημαντικό να μπουν στην έκθεση της ΛΥΠΕ. Ε, το ένα αφορά τη διαφάνεια. Νομίζω ότι η διαφάνεια είναι ένας μεγάλος βασικός παράγοντας ε, στον 21ο αιώνα για όλα όσα σημαίνει και λόγω όλων όσων σημαίνει η λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση και τις ε, ευκαιρίες που μας δίνει η τεχνολογία για να φτιάξουμε μια πιο ε, συμμετοχική δημοκρατία. Ε, ούτως ώστε να την έχουν όλοι. Στα δάχτυλα όλων. Νομίζω ότι η διαφάνεια είναι μία από τις αρχές που προστατεύει τη δημοκρατία από τη διαφθορά και τις ε, καταχρήσει. Ε, δεν νομίζω ότι αναφέρεται επαρκώ. Κάνω μια αναφορά επίσης στο ότι η πρωτοβουλία των πολιτών, τη συζητήσαμε προηγουμένως ε, με τον κύριο Σέφλινγκ, ε, είναι από τα βασικά στοιχεία που βελτιώνει την λειτουργία των δημοκρατιών μας και τέλος μια αναφορά στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Θέλω να το υπενθυμίσω γιατί στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι που δεν μπορούν να ψηφίσουν στι ευρωπαϊκέ εκλογέ. Πολλοί Ευρωπαίοι που επειδή δεν είναι στη χώρα του, όταν λαμβάνουν χώρα οι ευρωπαϊκέ εκλογέ, δεν ψηφίζουν. Έτσι και αυτό είναι θεμελιώδε δικαίωμα. Το δικαίωμα του να ψηφίζει. Ε, και παραβιάζεται δυστυχώ λόγω των εθνικών νομοθεσιών, που είναι ασύμβατε μεταξύ του και παράλογε. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία έβαλα. Επιτρέψτε να σας πω ότι η έκθεση Λίμπε, κατά την άποψή μου, ε, χρειάζεται έναν σημαντικό εμπλουτισμό. Ίσως με την ιδέα ότι δεν πρέπει να αναφέρουμε, να μπαίνουμε σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε ε, σε ό,τι αυτά τα προβλήματα, αλλά έτσι χάνουμε και έτσι επιρροή και σημασία. Να σα υπενθυμίσω επίση ότι Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει μια αιτήσια έκθεση για το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν όμω αναλύουμε τον εαυτό μα, όταν αναλύουμε τις εσωτερικές μας δυσκολίες, δεν θέλουμε να αγγίξουμε διάφορα πράγματα. Έτσι. Την, τα εσωτερικά θέματα ε, κάποιας χώρας. Ε, προσκρούμε στις ιδεολογίες κάποιων πολιτικών ομάδων, ομάδων πούμε, ή κομμάτων κτλ. Ε, πρέπει να είμαστε νομίζω όμως πιο επικριτικοί απέναντι στη δική μας την κατάσταση. Γιατί αλλιώς χάνουμε την επιρροή μας, την δύναμή μας, την ισχύ μας κτλ. Τέλος πάντων, ε, θα ακούσω τα σχόλιά σας και τις τροπολογίες με μεγάλο ε, ενδιαφέρον και πιστεύω ότι έτσι θα βελτιώσουμε και το κείμενο που παρουσίασα. Ευχαριστούμε. Στο Μάγκον Σάλες, για τους θα μιλήσετε ε, για λογαριασμό του. Καλώς. Ε, ναι, δεν μπορώ να μιλήσω άμεσα ε, ε, για λογαριασμό του, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς θα σας έλεγε, αλλά νομίζω ε, πως θα είχε δικές του τροπολογίες. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή και πράγματι το να θέσουμε εδώ τις, τα θεμελιώδη δικαιώματα στο επίκεντρο. Δηλαδή, ο κύριος Γουαρέκη μπορεί να μην συμφωνήσει με αυτό που θα πω, αλλά ε, το δημοκρατικό σύστημα σήμερα στην Ευρώπη είναι λιγότερο πολιτικό από ότι ήταν 30 ή 40 χρόνια πριν. Δηλαδή η πολιτική ισχύ έχει κατακαιρματιστεί, έχει δηλαδή μεταφερθεί σε μία σειρά από διαφορετικούς τομείς όπου οι πολίτες ως με την ιδιότητα του πολίτη δεν, έχουν, ε, δεν μπορούν να ασκήσουν μεγάλη επιρροή. Ναι, εντάξει, οι κυβερνητικές οργανώσεις εδώ ε, παίζουν έναν ε, ρόλο, αλλά αυτό είναι εκείνο που ε, περιορίζεται στο, σε αυτόν δηλαδή που δίνεται στου ίδιου του πολίτε. Άρα λοιπόν οι πολιτικέ αποφάσει πολύ συχνά γίνεται, γίνονται σε επίπεδο δικαστικών αρχών, το οποίο μερικέ φορέ είναι θεμητό, αλλά κάποιε άλλε όχι. Εν πάση περιπτώσει εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι εκεί ε, η χρειά που θα πρέπει να δώσουμε είναι ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να συνεχίσει να ξαναβρίσκει, να επανα ε, φέρει ε, στην ιστορροπία ιστοροπία ε, την κατάσταση όπως δηλαδή αυτή διαταράσσεται συνεχώς από τις εξελίξεις. Έχω να θέσω ένα ερώτημα τώρα στον κύριο Χαρόγγι. Όταν κάνετε αναφορά στις μειονότητες ήσασταν πολύ προσεκτικός προκειμένου ε, να μην διευκρινίζεται περαιτέρω. Δηλαδή μιλάτε και για ε, εθνικού γλωσσικού χαρακτήρα μειονότητες ε, και από εκεί και μετά τι θέλετε να κάνετε σε σχέση με τις νέες μειονότητες που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση. Για παράδειγμα η παλαιά εργατική τάξη η οποία ουσιαστικά ουσιαστικά βγαίνει από την αγορά σε διάφορα συμμετοχή μου Ε, και αυτό είναι το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω σε εσά. Δηλαδή, τι συμβαίνει με αυτέ τι νέε μειονότητε. Για την άλλη, λοιπόν, συγκητή. Ποιο είναι. Ευχαριστώ κυρία μου. Αυτή τη φορά είμαι εγώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή που μας εισήγαγε σε μια συζήτηση πραγματικά ενδιαφέρουσα. Μια φορά ακόμη ε, διαπιστώνουμε το χάσμα που χωρίζει από τη μία πλευρά την ανάγκη σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και από την άλλη πλευρά των περιορισμένων μέσων που συχνά έχουμε στη διάθεσή μας για να επιβάλλουμε κυρώσεις στις παραβιώσεις αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι αν κάνουμε μία απογραφή επιχειρημάτων για να τροποποιήσουμε τις συνθήκες. Η έκθεσή σας θα ήταν μια σημαντική συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση. Εξηγώ τι εννοώ. Ας πάρουμε τις συνθήκες που επιβάλλουμε στα κράτη όταν θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη συνθήκη της Κομπεχάης. Αναφέρεστε σε αυτήν είναι, ανήκει στην πρώτη κατηγορία κριτηρίων η συνθήκη της Κοπεχάγης, είναι τα πολιτικά κριτήρια που αφορούν και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μια χώρα η οποία δεν σέβεται σήμερα την ελευθερία των ΜΜΕ, τι μέσα έχουμε για να επιβάλλουμε κυρώσεις. Διαπιστώνουμε αδυναμία σε σχέση με τις συνθήκες όπως εφαρμόζονται. Η Κομισιόν είναι καταδικασμένη να περιοριστεί στον πολύ στενό τομέα της εφαρμογής του, της νομοθεσίας. Ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν έχει ας πούμε επικυρωθεί ή εφαρμοστεί σωστά από την εν λόγω χώρα. Η Κομισιόν πρέπει να παρέμβει αλλά δεν έχει τίποτα να αντιπαραθέσει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε επιτέλους τα μέσα εφαρμογής ε, όπως όταν επιβάλλουμε όρους για τις συνεκβανών, όρους για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά είναι παραπάνω από βέβαιο ότι μεσοπρόθεσμα θα χρειαστεί να μετροποποιήσουμε τις συνθήκες. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Ας πάρουμε το οργανισμό της Βιέννης για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εκτός αν κάνω λάθος, πρόκειται για ένα όργανο το οποίο είναι στη διάθεση της Κομισιόν. Όμως αυτός ο οργανισμός δεν μπορεί να αυτό ασχοληθεί με ένα θέμα και να το φέρει στο προσκήνιο. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα από τη στιγμή που διαπιστώνεται στην παρακολούθηση που γίνεται της εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που διαπιστώνει λέω μια παραβίαση θα πρέπει να μπορεί να αυτό αν αποφασίσει από μόνη της να ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση, να τη φέρει στο προσκήνιο και από το γεγονός ότι δεν έχει το δικαίωμα αυτό να αναλάβει πρωτοβουλία σε αυτό το τομέα και να το φέρει, φέρει θέματα στη δημοσιότητα, ε, συνεπάγεται ανεπάρκεια μέσων. Και ακριβώς αυτή τη δημόσια συζήτηση πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε μια πολιτική δύναμη και μπορούμε να πιέσουμε τα πράγματα καλύτερα αν ο οργανισμός που ανέφερα στη Βιέννη μπορούσε να προχωρήσει αυτόνομα. Ευχαριστώ. Η Μπάρμπα Σπινέλη τώρα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ θερμά τον εισηγητή για την γνωμοδότηση. Τον κύριο Χαουρέγγι Ατόντο για τη θαυμάσια γνωμοδότηση. Καταρχάς, μιλάτε για την προσχώρηση στη σύμβαση ε, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω της απόφασης του δικαστηρίου. Πρέπει να είμαστε πολύ απαιτητικοί σε αυτό και να ζητήσουμε να, επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσει στο στομότερο δυνατόν, να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει στο στομότερο δυνατόν. Να μην υπενθυμίσουμε απλώ την δέσμευση που έχουμε λάβει για προσχώρηση, αλλά να πιέσουμε για μια ε, γρήγορη επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, κάτι που συνδέεται με το πρώτο, είναι οι επιπτώσεις της κρίσης και της θεραπείας ε, για την καταπολέμηση της κρίσης στα θεμελιώδη δικαιώματα και στα κοινωνικά δικαιώματα. Τι κάνουμε. Καταρχάς, πρέπει να προσχωρήσουμε στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δεύτερον, να προσχωρήσουμε στην ε, Χάρτα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και να σεβαστούμε τη Χάρτα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό για να αντιμετωπίσουμε ε, τις επιπτώσεις της κρίσης στα θεμελιώδη δικαιώματα, τις αρνητικές επιπτώσεις. Να σας υπενθυμίσω κάτι που είναι πολύ λεπτό κατά την άποψή μου, τις ε, συμφωνίες που δεν είναι κοινοτικέ, είναι διεθνείς, όπως παραδείγματος χάρη το Fiscal Compact, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Τι σχέση έχουν αυτές οι συμφωνίες και το Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου. Με το Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου, τι σχέση υπάρχει. Και με την ε, Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν διαφορετικές και αντιφατικές μεταξύ τους ερμηνείες της Κομισιόν. Ο Επίτροπος Κατάινεν, η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου ας πούμε, αναστέλλεται τροποντινά όταν εφαρμόζεται παραδείγματο χάρη το Fiscal Compact, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, στην Ελλάδα. Οι πολιτικές κατά της κρίσης τη συμφωνεί το κράτος με τους πιστωτέ του. Άρα δεν επικυρώνονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Άρα δεν ισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο Τίμερμαν όμω λέει ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο, το ευρωπαϊκό rule of law, το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου ποτέ δεν αναστέλλεται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επουδενή. Υπάρχει σαφώς λοιπόν μια διαφορετική ερμηνεία. Ένα άλλο σημείο που μου φαίνεται σημαντικό είναι το εισόδημα των πολιτών, που είναι θεμελιώδες δικαιώματα και πρέπει να το, ε, και πρέπει να το υπενθυμίσουμε. Είναι σημαντικό τη στιγμή που υπάρχει μια απογοήτευση από του, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με αυτό το, το εισόδημα υπάρχουν και τα ατομικά δικαιώματα και τα συλλογικά δικαιώματα. Να μην τα ξεχνάμε. Παραδείγματο χάρη, ε, το να έχεις πρόσβαση στο νερό. Ε, νερό που να μην κατέχεται από ιδιωτικέ εταιρείε. Το, το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Θα ήθελα να μου πείτε τη την γνώμη σας για αυτό το θέμα. Τελευταίος ομιλητής είναι ο κ. Καστάλντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ, συνάδελφε, για τη δουλειά σας. Σε την, για τη δουλειά που κάνατε με αυτή την ε, γνωμοδότηση και τώρα θα μιλήσω Ιταλικά, γιατί τα πρώτα ήταν Ισπανικά. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα-δύο σημεία. Το σημείο 3, το οποίο μιλάει για, την καρδιά της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή που πρέπει να είναι η καρδιά κανονικά, που, που είναι η κοινωνική Ευρώπη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία της Ένωσης συνολικά συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής να εφαρμόζεται σύμφωνα με το χάρτη Μελιωδών δικαιωμάτων. Η ερώτηση της κυρία Πινέλη είναι κέρια για αυτό το σημείο. Τι σχέση υπάρχει με τις ε, συνθήκες που υποτίθεται αυτές ε, διέπουν, ε, καθορίζουν το δίκαιο της Ένωσης. Αλλά μην ξεχνάμε και όλες τις υπόλοιπες συμφωνίες που έχουμε, τα προγράμματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι η σχέση όλων αυτών. Θα πρέπει η δράση να είναι ε, αναλογική με τους σκοπούς που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Και οι πολιτικές λιτότητας μέχρι στιγμής που υιοθετήθηκαν για να αντιμετωπιστεί η κρίση, κατά την προσωπική μου γνώμη, αλλά και κάτι τη πολλών. Δεν νομίζω ότι εφαρμόστηκαν ε, σωστά με βάση τις αρχές μας, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές μας, ε, με βάση τις αρχές στις οποίες ιδρύθηκε η Ένωση με βάση τις ε, θεμελιώδεις αξίες μας. Και εδώ θα πρέπει να, να υπάρξει και μια διασύνδεση με τη γνωμοδότηση για την οποία σας μίλησα σήμερα το πρωί, όπου ο έλεγχος θα πρέπει να γίνει όχι μόνο κατά την εφαρμογή, αλλά και κατά την υποδοχή, την εσωμάτωση δηλαδή, στα στην νομοθεσία των κρατών μελών. Και αυτό θα πρέπει να αναφερθεί. Και θα είναι μια θαυμάσια πηξίδα ε, θα μπορούσαμε να το δώσουμε ως εργαλείο στους εθνικούς βουλευτές για να αποτρέψουμε το να υπάρχουν ασυμβατότητες πριν καν λάβουν χώρα, δηλαδή να τις αποτρέψουμε. Μου άρεσε αυτό που είπατε για την ε, δημοκρατία ως ε, προστασία των μειονοτήτων. Γιατί και αυτό είναι η δημοκρατία. Συχνά ε, στις διάφορες, στα διάφορα κοινοβούλια ε, θεωρούμε καμιά φορά ότι η δημοκρατία για των πολλών. Όχι, προστασία των μειονοτήτων αντίθετα είναι δημοκρατία ε, στα πλαίσια του Κοινοβουλίου αλλά και στο εσωτερικό μιας χώρας, ε, στην κοινωνία των πολιτών κτλ. Το τελευταίο, στο σημείο 6, εκεί που γίνεται λόγος για διάφορα στοιχεία. Νομίζω ότι πρέπει να, εδώ να κάνουμε μια τροπολογία για το σημείο αυτό 6 και να ζητήσουμε μία δέσμευση για να ε, ο, ακυρώσουμε όλα τα οικονομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που αναφέρονται πολύ σωστά, αναφέρθηκαν πολύ σωστά από τον κύριο Σέπλικ πριν, που ε, καθιστούν πάρα πολύ δύσκολη την προώθηση της πρωτοβουλίας των πολιτών, ε, η οποία συνδέεται τόσο πολύ με την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας. Εάν δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία και κυρώσει ενδεχομένω αν χρειαστεί, όχι μόνο πρόθεση αλλά και κυρώσει, για να εξασφαλίσουμε την, τα θεμελιώδη δικαιώματά μα, μπορεί στο μέλλον να υποσκαθούν ή να παραμείνουν γράμμα κενό περιεχομένου. Να παραμείνει στα χαρτιά δηλαδή, αλλά που δεν έχει καμία πρακτική επίπτωση, ας πούμε, στην καθημερινότητα των πολιτών. Ε, Ράμον Έχετε να αντιδράσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Οι παρατηρήσεις των συναδέλφων όλες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ήταν επίσης και στη συζήτηση που κάναμε πριν ετοιμάσω αυτή την γνωμοδότηση. Όλε οι παρατηρήσει δηλαδή, που άκουσα μέχρι στιγμή και πριν και τώρα ήταν χρήσιμε. Σε ό,τι αφορά του μηχανισμού για την αποκατάσταση των παραβιασμένων, για να το πω έτσι, ε, δικαιωμάτων. Νομίζω ότι αυτή ήταν η έκφρασή σας. Τι να σας πω. Νομίζω ότι υπάρχει ο μηχανισμός. Να σας υπενθυμίσω ότι το άρθρο 2 της συνθήκης λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δημοκρατία κτλ. Και στο 7, στο άρθρο 7 λέμε ότι, για, ότι χρειάζεται για την τροποποίηση το 1 τρίτο των ε, μελών. Και στο Συμβούλιο με πλειοψηφία τετάρτων, των 4 πέμπτων. Ε, μπορούμε να διαπιστώσουμε την ε, ύπαρξη ενός σαφούς κινδύνου παραβίασης από πλευράς ενός κράτους Επομένως, αυτό που μας είπατε, ότι απαιτούμε πολλά από τα κράτη για να ε, ενταχθούν αρχές της Κοπενχάης και μετά αυτή τη στιγμή μπουν τα κράτη, ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει ουσιαστικά. Ε, αυτό με απασχολεί πάρα πολύ, με ανησυχεί πάρα πολύ. Συμβαίνει αυτό. Η εφαρμογή αυτού του μηχανισμού όμως πρέπει να διαπιστώσουμε ότι πολιτικά ε, πού οδηγεί. Ε, στην πραγματικότητα ποτέ δεν εφαρμόστηκε είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Και αυτό η Κομισιόν έφτιαξε αυτή τη διαδικασία και υπ' αυτή την έννοια να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε και ένα έγγραφο που μόλις ανέκρινε η Κομισιόν, το 2014 συγκεκριμένα, το οποίο είναι μία ανακοίνωση. 2014, 11 Μαρτίου του 2014 και που την όλη διαδικασία, αναφέρει τη διαδικασία ούτως ώστε η Ένωση να αποκτήσει μηχανισμούς ελέγχου κατά των παραβιάσεων από τα κράτη-μέλη. Η συγγήτρια του, της ΛΥΜΠΕ, η κυρία Φεράρα, στην έκθεσή της, λέει ότι ο μηχανισμός της φαίνεται ανεπαρκής και αναφέρει και μία σειρά στοιχείων που μπορούν να βελτιώσουν το μηχανισμό. Αυτά υπάρχουν στην έκθεση. Είναι βασικό στοιχείο αυτή τη συζήτηση. Γιατί σίγουρα θα πρέπει να δούμε εάν τα εργαλεία που αναφέρουν οι συνθήκες, εάν παρόλα αυτά υπάρχει δυνατότητα, εάν ένα κράτο ε, προβεί σε κάποια παραβίαση, να μπορέσουμε να το ανακαλέσουμε στην τάξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολιτικά είναι πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να μιλήσω για καμία χώρα, να υποδείξω καμία χώρα. Ας πούμε ότι μια χώρα, ας πούμε, με αυτή τη διαδικασία και αφού, κάνει μια έκθεση προηγουμένως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκινάει, ας πούμε, μια διαδικασία επί παραβάση, ας πούμε. Υπάρχει αυτή η διαδικασία. Οι, οι μειονότητες που μου λέει ο κ. Σόπλιν, για μένα όλες οι μειονότητες είναι εθνικογλωσσικές, Φερρυπίν. Δεν είναι οι γλώσσες που έχουν τα δικαιώματα, αλλά τα άτομα που μιλάνε αυτές τις ε, γλώσσες, Φερρυπίν. Μειονότητες είναι και αυτές. Όταν ένα σύνολο ανθρώπων μιλάει μία γλώσσα, εάν αυτή η γλώσσα δεν προστατεύεται, τότε να ένα πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιου τύπου πολλά προβλήματα στην Ευρώπη. Υπάρχουν μεγάλες μειονότητε που δεν μπορούν να εκφραστούν στη γλώσσα τους σε πολλές χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Και αυτό είναι πρόβλημα, σαφέστατα. Αυτό είναι το σχόλιο που σας έκανα λιγάκι προηγουμένως. Ε, ας κάνουμε μία έκθεση αναχώρα, χώρα προς χώρα. Τι γίνεται σε κάθε χώρα. Γιατί όχι. Δεν είναι και τόσο απίθανη ιδέα. Επίσης, αυτό που είπε η κυρία Σπινέλη και ο κύριος Καστάλντο. Τι γίνεται με όλο αυτό που φτιάξαμε, που χτίσαμε από το 1950 μέχρι το 80, 90 κτλ. Ε, αυτό το κοινωνικό εργατικό πλαίσιο. Ε, φτιάξαμε ένα ολόκληρο δίκαιο, έτσι που, προστατεύει συγγνώμη, τον εργάτη απέναντι στην επιχείρηση κτλ. Τι γίνεται με τη συστηματική ε, υποτίμηση αυτού του πλαισίου, την υπόσκαψή του. Τι γίνεται. Υπάρχει ένα σαφέστατο πρόβλημα εδώ. Σε σχέση με αυτό που μου έλεγε η κυρία Σπινέλη για το νερό, ας πούμε. Τι απάντηση δίνεται γι' αυτό, για αυτό το πρόβλημα. Ίσως θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι, να φτιάξουμε μια νέα ε, κοινωνικο-εργατική ε, τάξη, ένα νέο εργατικό κοινωνικό πλαίσιο για τον νέο κόσμο, για την νέα εποχή ας πούμε. Η εργατική τάξη οι προλετάροι απαιτούν, χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία ίσως. Τι αναφορές υπάρχουν. Για μένα υπάρχουν δύο. Ε, η κοινωνική χάρτα που δεν, είναι, είχε εγκριθεί από όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλειοψηφία ναι. Και δεν έχει ενσωματωθεί ε, και δεν έχει γίνει βασικό κείμενο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, αυτό το λέμε σε αυτή την έκθεση. Δεν υπήρχε στην έκθεση τη ΛΥΜΠΕ. Εγώ το έβαλα στο δικό μα κείμενο. Λέμε ότι η κοινωνική, η ε, κοινωνική χάρτα θα πρέπει να είναι σημείο αναφορά ε, για να υπάρχει ένα ελάχιστο σεβασμό σε αυτό που λέμε ας πούμε κοινωνικοεργατική ας πούμε αξιοπρέπεια. Έπειτα δεύτερο στοιχείο αναφορά. είναι οι συλλογικέ συμβάσει. Ο διάλογο αυτό, ο κοινωνικό και εργατικό διάλογο, για να οικοδομηθεί αυτό ο κόσμο, αυτό το πλαίσιο που σα ε, έλεγα. Υπάρχει παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όταν εφαρμόζεται το σύμφωνο σταθερότητα. Ναι, χρήζει ερμηνεία σίγουρα αυτό. Σίγουρα. Ενδεχομένως η εφαρμογή μιας ε, υπερβολικής ε, λιτότητας θίγει δικαιώματα. Από την άλλη μεριά, οι μακροοικονομικές πολιτικές απαιτούν μέτρα. Έτσι δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση όμως. Ε, αλλά και το ένα είναι δικαίωμα και το άλλο είναι δικαίωμα. Στην τελική δηλαδή φάση υπάρχουν νομικοί κανόνες και πρέπει να τους εφαρμόσουμε. Αυτό που λέμε εδώ, κυρία Σπινέλη, δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα από το να πούμε ότι η εφαρμογή των μακροοικονομικών πολιτικών όταν γίνονται εφαρμόζονται ως προσαρμογές σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ε, παραβιάζουν ας πούμε τα εργατικά ε, δικαιώματα και τα κοινωνικά δικαιώματα που είναι θεσπισμένα και καθιερωμένα παραδείγματο χάρη ε, ιδιωτικοποίηση του νερού σίγουρα παραβιάζει ε, το δικαίωμα στο νερό. Υπάρχουν νομικέ ερμηνείε που λένε όμω και ερμηνεύουν και καταφέρουν να ανασκευάσουν αυτή την ιδέα και λένε ότι δεν παραβιάζουν αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα. Γιατί μπορεί μια δημόσια υπηρεσία να μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί ε, υπό τον όρο ότι γίνονται σεβαστέ κάποιε προποθέσει. Είναι πάρα πολύ λεπτές συζητήσει και δεν μπορούμε να τι επιλύσουμε εδώ πέρα σε αυτό το κείμενο. Θέλω να σα πω ότι το πολύ πολύ που μπορούμε να κάνουμε στην ΑΦΚΟ είναι να εκδώσουμε μία γνωμοδότηση αναφερόμενη σε αυτά τα στοιχεία που σας είπα και σας προσκαλώ εσάς να υποβάλλετε τις ε, τροπολογίες που θεωρείτε απαραίτητες και σας ε, διαβεβαιώ ότι θα φτιάξουμε μία γνωμοδότηση που εμπλουτίζει την έκθεση της κυρίας Φεράρα της ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ. Έχω μία δύσκολη κατάσταση μάλλον. Γι' αυτό και το κείμενο απεστάλλει πριν από δύο εβδομάδες στους κοιόδης και στους πολιτικούς συμβούλους. Διότι το μέγιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι ε, η προθεσμία τροπολογιών να είναι αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται, 20 Απριλίου, 4 μετά μεσημβρίας. Μόνο έτσι μπορούμε να αποστείλουμε τη γνωμοδότηση εγκαίρως στη Λίμπε πρωτού ψηφίσουμε. Ελπίζω λοιπόν ότι θα το δεχτείτε, θα το δεχτείτε αυτό και κλείνω αυτό το θέμα συζήτησης. Έχουμε ακόμη δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα διάφορα δεν έχουμε τίποτα σε αυτό, κάτω από αυτό και θα ήθελα να σας ενημερώσω αυτόν τον δεύτερο, 5 Μαΐου έχουμε μια, την επόμενη μας συνεδρίαση και σας ευχαριστώ για όλα. Γεια σας.